Γεια σας, κύριε Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως είπαμε, θα αρχίσουμε στις 3 και θα συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών με μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων. δύναμη του άρθρου 51 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Αυτό το που θέλουμε να κάνουμε είναι να συζητήσουμε το πρόγραμμα για την πολιτική της δικαιοσύνης 2014-2020. Και να ακούσουμε την εισήγηση της κυρίας Παρασκευή Μισού, που είναι η Διευθύντρια για τα θέματα αστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνεχεία δε, πρόκειται Παρασκευή Μίχου. Παρασκευή Μίχου, ζητήσει συγγνώμη τη Θα ακολουθήσει συζήτηση επί αυτού του προγράμματο για την δικαιοσύνη στα πλαίσια του πολιετού δημοσιονομικού χρηματοδοτικού πλαισίου μέχρι το 2020. Να δούμε πώ θα πρικοδοτηθούν οι δραστηριότητε για αυτή την ε, ευρωπαϊκή, τον ευρωπαϊκό χώρο Δικαιοσύνη. Πρόκειται ακριβώ για το πρόγραμμα 2014-2020, το οποίο πρόκειται να διαδεχθεί Τρία υπάρχουν τα προγράμματα τα οποία τώρα, τώρα βρίσκονται εν εξελίξη για, για αστική δικαιοσύνη, ποινική δικαιοσύνη, τρίτον καταπολέμηση ε, ναρκωτικών και τέταρτον ε, πρόγραμμα πληροφόρηση και ενημέρωση. Οπότε θα δούμε πώ αυτά τα τρία πρόκειται να ενοποιηθούν ει ένα και έτσι να έχουμε ένα μέσο πολιτική και επίση να μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποια προσέγγιση χρηματοδοτική για την πολιτική δικαιοσύνη και να έχουμε πιο ορθολογικό τρόπο κατανομή των ε, κονδυλίων για κάποια οριζόντια ζητήματα μεταξύ των οποίων είναι και η εκπαίδευση των δικαστικών. Οπότε εμεί είμαστε συνυπεύθυνοι στι αρμόδιε επιτροπέ του Κοινοβούλου, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και η Επιτροπή Νομικών Ελευθεριών και στα πλαίσια του άρθρου 51 εργαζόμαστε. Θα έχουμε το επομένω την ε, εισήγηση, την παρουσίαση από την κυρία Μίχου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια οι εισηγητέ, ο κύριο Φίλιπ Κλάι και για την Νομική Επιτροπή συγγνώμη, ο πρώτος για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθερών και για την Νομική Επιτροπή, ε, κ. Μπερλιγκουέρ, δεν λέει ο πρόεδρο. Τώρα, τώρα, τώρα στρεφόμαστε στον κ. Μπερλιγκουέρ, που είναι ο αντιπρόεδρο τη Νομική Επιτροπή, ο οποίο επίση πρόκειται να συμπροεδρεύσει τη ε, συνάντησή μα. Ε, πριν λάβει το λόγο η κυρία Μίχου. Είναι. Λάβανε τώρα το λόγο ο κ. Μπερλιγκουέρ. Δεν θέλω να εκμεταλλευτώ, να, να διασπαθήσω, να αλλώσω το χρόνο σας. Πάντως και εγώ ήθελα να σας πω δύο λόγια, μια που είμαι και εγώ εισηγητής. Ε, θα σας τα πω σε λίγο. Αυτό το οποίο θέλω προς το παρόν να τονίσω είναι ε, το πόσο σημαντική είναι η υπόθεση αυτή την οποία σήμερα συζητούμε, αυτό το πρόγραμμα για την δικαιοσύνη, ε, να δούμε πώς θα έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών μας, των συναρμοδίων και προσέξτε, δεν είναι η πρώτη φορά Πού συνεργαζόμεθα. Δεν είναι η Δεν, δεν είναι, γιατί έχουμε ακριβώς αυτές τις ε, ε κοινέ αρμοδιότητες, τα θέματα πολιτική, πολι... αστικού δικαίου, ποινικού δικαίου. Και ε, γι' αυτό το λόγο και κάνουμε αυτή την κοινή συνάντηση, ε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται, τα βασικά στοιχεία αυτού του προγράμματος, αυτού του διαδήματος. Οπότε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ακριβώ επιτελούμε το έργο μα χέρι-χέρι. Λέγει ο Σπέρλινγκουερ. Πρόεδρο Λόπε Αγγελέα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σπέρλινγκουερ και τώρα πρόκειται να ακούσουμε την παρουσίαση τη Διευθυντρία Αστικού Δικαίου ε, τη κυρία Μίχου. Mr. Solskov Lind, representing the Danish presidency. Κατόπιν θα ακούσουμε και εκπρόσωπο της ε, Δανέζικης Προεδρίας. Πρώτα πρώτα, η κυρία Μίχου θα έχει το λόγο. Βρίσκεται εδώ. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Κυρία Μίχου, έχετε το λόγο. Time. Good afternoon. Ήρθα, στην ώρα μου. Καλησπέρα όλοι, λέει η κυρία Μίχου. Καλησπέρα όλοι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε και που μα δώσατε την ευκαιρία να σα ε, παρουσιάσουμε αυτά τα προγράμματα. Στι 15 ε, Νοεμβρίου ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την πρόταση, ούτω ώστε να εγκριθεί, για να συγκροτηθεί αυτό το πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020. Τα άλλα προγράμματα τα οποία επίση έχουμε προτείνει αφορούν τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Αυτό όμω όταν έρθει η ώρα σε κάποια άλλη συνάντηση, όταν χρειάζεται, θα σα το παρουσιάσω και σε αυτή τη συνάντηση. Γιατί τέλο πάντων το ένα πρόγραμμα επικαλείται κάποιο τρόπο με το άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για του επιλέξιμου, για όσου θα καλυφθούν στο μέλλον, ε, για όσου τέλο πάντων εμπλέκονται. Ε, τα προγράμματα αυτά πρέπει να ξέρετε επομένω όλοι ότι έχουν παρόμοια δομή. Όλα αφορούν κάποια εύρυθμη λειτουργία τη δικαιοσύνη, εύρυθμη λειτουργία τομέα τη δικαιοσύνη. Οπότε έχουμε αυτό το προτινόμενο πρόγραμμα όπου έχουμε συγχώνευση αυτών των τριών προεπαξάντων προγραμμάτων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει μεγάλη πρικοδότηση. Μιλούμε για λιγότερο από το 0,1% της, ε, του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως παρόλα αυτά βοηθά πάρα πολύ σημαντικά ε, την λειτουργία των δικαϊκών συστημάτων των κρατών μελών και μια που πρόκειται για μια συγκυρία οικονομικής ε, κρίσης ε, θα πρέπει να διστακτικοί ή στο να αναλώνουμε το χρήμα των φορολογουμένων όπου δεν υπάρχει προστεμένη αξία. Και όταν λέμε για κοινωτική προστεμένη αξία σημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός προπολισμός θα πρέπει να ε, λειτουργεί στην περίπτωση όπου δεν μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν οι περιφέρειες, τα κράτη-μέλη και μόνο εκεί όπου μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους ε, Ευρωπαίους. Τώρα, εμείς ε, είμαι θα υπέρ αυτού του προγράμματος επομένως για να δούμε πώς θα δημιουργηθεί, ολοκληρωθεί αυτός ο χώρος δικαιοσύνης, ε, να δούμε πώς θα προωθήσουμε κάποιες λύσεις σε θέματα δικονομικά και αστικού δικαίου, πώς θα είναι τα... η δικαιοσύνη των κρατών μελών πιο αποτελεσματική, πώς θα το περιμένουμε αυτό με το να έχουμε κάποιο είδους χρηματοδότηση ε, κατάρτισης και υποστήριξη της δράσης των εμπλεκομένων στην δικαιοδική διαδικασία και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο στην, για, για τις ποινικές και για αστικέ υποθέσεις. Η εκπαίδευση των δικαστών τονίστηκε από το ψήφισμά σας που ξεκίνησε με αφορμή δηλαδή στη δική μας ανακοίνωση για το πρόγραμμα τη Στοχόλμη. Υπήρχε ότι αυτό είναι μια προϋπόθεση ούτω ώστε να υπάρχει μια τέτοια ενιαία ευρωπαϊκή νομική κουλτούρα. Οπότε και να διευκολύνουμε τώρα την προσβασιμότητα στην πληροφόρηση και την ανταλλαγή δεδομένων στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να δούμε πώ η ερμοδότηση των προγραμμάτων πρόκειται να μα βοηθήσει να, να έχουμε κάποιο είδου ε, εργαλεία πολιτική τα οποία να ε, λειτουργούν διαλειτουργικά αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και σε, θα έχουμε επομένω κάποιο είδου ε, πύλε ηλεκτρονικέ ε, όπως το e-justice ε, και έτσι να μπορούν οι πολίτες να, να για το τι είδους προσβασιμότητα, τι είδους ε, αρρωγή υπάρχει νομική, ε, τι, έχουμε, τι, τι μητρώα έχουμε, όπως ας πούμε τα, τα, τα πτωχευτικά μητρώα, όπως ας πούμε τα κτηματολόγια κλπ. Και έτσι να έχουμε και κάποιο είδους διασυνοριακή δράση των ε, επιχειρήσεων σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Επίση, αυτό το πρόγραμμα να καλύψουμε και κατανοήσει των ναρκωτικών και θέλουμε να βοηθήσουμε τη συνεργασία των μελών ε, για την καταπολέμηση τη λαθρεμπορία ναρκωτικών και πρόκειται για ένα τομέα όπου ο Ευρωπαϊκό Νομοθέτη μπορεί να θεσπίσει κάποιου ελάχιστου κανόνε όσον αφορά τα σχετικά εγκλήματα, εγκλήματα επιθέσματα κλπ. Και σα παραμένω στο άρθρο 83. Αν τώρα κάτσετε και συγκρίνετε τι ισχύει σήμερα όσον αφορά το ενημερωτικό πρόγραμμα για τα ναρκωτικά, το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με θέματα υγεία, εμεί αλλάξαμε ρότα τελείω. Και τώρα ο σκοπό μα είναι να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη, μεγαλύτερη επιρροή στο γίνεστε σε αυτόν τον τομέα. Να σου πω τώρα μερικέ λεπτομέρειε, όσον αφορά την προσέγγιση μας ε, έχουμε Επομένως το υφητήσαν μια τελείως καινούργια οπτική γωνία και παρά το ότι είδαμε, διαπιστώσαμε τι γίνεται με τους ευλογωμένους, ε, με τους καλυπτόμενους ε, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των σημερινών προγραμμάτων ε, για, για τους ελέξιμους μας είπαν παρατηρήσεις και, και για τα υπέρ και για τα κατά αυτών των προγραμμάτων. Οπότε επί τη βάση αυτή, αυτού του προγράμματο προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε αυτά τα κενά και αυτό ιδίω όσον αφορά την προσθέμενη αξία και τη διαχείριση. για να δούμε επομένως να τελικά θα προεκοδοτηθούν αυτά τα προγράμματα και ε, προσπαθήσαμε μέσα να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας είπαν οι μπλεκόμενοι. Θα πρέπει επομένω κανεί να έχει διαφορετική νοοτροπία όταν κάθεται να αναλύσει τι σχετικέ ε, προτάσει και εκείνε τι οποίε εμεί ε, το προτείνουμε, γιατί υπάρχει εδώ πέρα μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα. Οι στόχοι μα είναι το να έχουμε αυτό το streamlining, την ένταξη δηλαδή των επιμέρους πολιτικών στις υπόλοιπες, να έχουμε κάποιο αποτελεσματικότητα, να έχουμε επιπτώσεις ουσιαστικές και θα συμφωνείτε ότι ε, δεν είναι πολύ δύσκολο κανείς να προβλέψει ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του 2020. Και για αυτό το λόγο και εμείς ε, δεν θέλησαμε να δούμε το θέμα πάρα πολύ στενά και επίσης ε, είπαμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια μεγαλύτερη ευελιξία σε το τι ισχύει σήμερα. Streamline και, και απλούστευση θα πει ότι τα προγράμματα τώρα ευθυγραμμίζονται με τον δημιουργικό κανονισμό. Ε, και αυτό γίνεται χωρίς να επαναλαμβάνονται οι σχετικές διατάξεις ε, όπου, υπάρχει κάποια διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ό,τι υπάρχει σήμερα, ό,τι προβλέπεται για δράση, για διαγωνισμούς, προμήθειες και όλα αυτά Ακόμα και αν ε, υπάρχουν και κάποιοι τομεί λειτουργία των προγραμμάτων που δεν έχουν τι προτάσει, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται πλέον να χρηματοδοτούμε κάποια δίκτυα. Επίσης, η επιλέξιμη δεν θα διάπονται από κάποιους περιορισμούς. Ποιοι δηλαδή θα λαμβάνουν χρηματοδότηση. Νομικά πρόσωπα, κρατικές αρχές, όλοι, όλοι δυνητικά μπορεί να είναι επιλέξιμοι για αυτή τη χρηματοδότηση. Επίσης, για να μην ευνοήσουμε κάποιους από τους επιλέξιμους, είπαμε ότι δεν πρόκειται να κατονομάσουμε κάποιο νομικό πρόσωπο, κάποια νομική οντότητα ή στην πρόταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποιο νομικό πρόσωπο, κάποιος φορέας ο οποίος ε, ε, ε, μπλέκεται και κατά σημαντικό τρόπο στις πολιτικές ένωσες ε, αποκλείεται από ε, το να γίνει επιλέξιμος. Και ε, τώρα που θα κάνουμε αυτή τη συγχώνευση των υπαρχόντων προγραμμάτων, αντί για εκείνα τώρα, για να διευκολύνουμε τη ζωή των χρηστών των εμπλεκομένων, έχουμε δύο προγράμματα. Και θα ε, διέπονται ψήφιες διατάξεις ακριβώς όπως και για, την, για το τομέα της δικαιοσύνης δεν θα έχουμε επόμενες ενιαίες διατάξει ε, διατάξεις αντί για, για τα έξι διαφορετικά τα διατάξεων που γίνουν σήμερα. Έχοντας αυτά επομένως υπόψη, αυτό που θα κάνουμε τώρα σήμερα είναι να έχουμε μια καρποφόρα συνεργασία με εμάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι να εξασφαλίσουμε το ότι αυτές οι προτάσεις θα εγκριθούν κατά τη διάρκεια του 2012 να <clears throat> έχουν αρχίσει οι επαφέ ε, με το Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και αν τυχόν έχετε τίποτα ερωτήσει να απαντήσω. Ευχαρίστω. Εμεί ευχαριστούμε, λέει ο κύριο Λόπε Αγγιλάρη. Ευχαριστούμε για την προσοχή σα και τώρα να ακούσουμε τι είχε να μα πει ο εκπρόσωπο τη Δανέργεια Προεδρία, ο κ. Σόλσκοφ Λίντ. Έχετε το λόγο, κύριε. Εσά ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι διαπραγματεύσει για την πρόταση αυτή μόλις ξεκίνησαν στο Συμβούλιο μια νέα ομάδα ad hoc δημιουργήθηκε με στόχο την διαπραγμάτευση των νέων προτάσεων στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και της δικαιοσύνης. Ο χρόνος βέβαια είναι σημαντικός παράγων στις διαπραγματεύσεις αυτές γιατί λήγουν τα προγράμματα χρηματοδότησης το 2013 και θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε έφθετο χρόνο τα νέα προγράμματα. Γι' αυτό ακριβώς η Προεδρία προωθεί το θέμα αυτό στο Συμβούλιο κατά προτεραιότητα. Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας ad hoc έδειξε ότι όλα τα κράτη-μέλη συμμερίζονται τις προδοκίες της Δανίας. Επί της ουσίας, η συζήτηση έδειξε ότι όλα τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν τις προσπάθειες απλούστευσης και ορθολογικοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της δικαιοσύνης. Η πρόταση της Επιτροπής στηρίζεται εμπολής από τα κράτη-μέλη σχετικά με τους στόχους και τις δράσεις. Περαιτέρω συζητήσεις βέβαια θα πρέπει να γίνουν στο Συμβούλιο και η Προεδρία περιμένει να συζητήσει το θέμα αυτό με πολύ ενδιαφέρον και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις πρώτες απόψεις του Κοινοβουλίου. Καλώς. Θα ξεκινήσει η συζήτηση. Θα περάσουμε πρώτα στον εισηγητή. Ή ε, μάλλον για μια στιγμή κύριε Κλάις, πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπερλίνγκουερ. Σαν συμπρόεδρος και μετά κύριε Κλάις θα επιστρέψουμε σε εσάς. Κύριε Μπερλιγκουέ, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία σκέψη που αφορά το πολιετές πρόγραμμα. Είμαι πεπισμένος ότι το πιο ουσιαστικό θέμα στον τομέα της πολιτικής και της δικαιοσύνης είναι η έλλειψη ισορροπίας που χαρακτηρίζει από τη μία μία θα έλεγα σημαντική νομοθετική παραγωγή είτε σε επίπεδο νομολογίας είτε σε επίπεδο νομοθετικό από πλευράς δικαστηρίων το πρώτο, από πλευράς Συμβουλίου και Κοινοβουλίου το δεύτερο και την διαφορά που χωρίζει αυτά τα αποτελέσματα από τον καθημερινό πολίτη της Ένωσης πολίτης, ο μεσαίος πολίτης, ο οποίος ζητά να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του και οι προσδοκίες του. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο μπροστά σε αυτό το σύνολο θα έλεγα των νομοθετικών προτάσεων. Έχουμε λοιπόν σε ένα σημαντικό βαθμό ένα πρόβλημα εφαρμογής των υπαρχουσών διατάξεων. Έχει δημιουργηθεί ο χώρος ο λεγόμενος Τζάι. Έχουμε προχωρήσει τώρα πια και στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Και μετά και από τις καινοτομίες που εισάγει η συνθήκη της Λισαβόνας, φαίνεται να υπάρχει μία ανάγκη από πλευράς της Ευρώπης και των μεμονωμένων κρατών μελών, που κινητοποιούνται μέσω της Ευρώπης, να θέσουν εν πολύ στο θέμα της εφαρμογής αυτών των μέτρων. Οι εθνικοί δικαστές και όχι μόνο τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αλλά και οι δικηγόροι σε εθνικό επίπεδο εισάγουν το ευρωπαϊκό δίκαιο στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων. Πιστεύω λοιπόν ότι μια πρώτη σκέψη την οποία θα πρέπει να εκφράσω μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η θεματολογία αυτή η οποία είναι παρούσα στο πολιετές πρόγραμμα θα πρέπει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο βάρος και θα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πολλαπλών φύσεων παρεμβάσεων για την επίτευξη του στόχου που θα επιτρέψει στους πολίτες να γνωρίσουν πρώτα τα δικαιώματά τους επί τη βάση του Ευρωπαϊκού Νομικού Συστήματος, γιατί περισσότεροι πολίτες δεν τα γνωρίζουν τα δικαιώματα αυτά. Και μετά να επιτρέψουν στους χρήστες του δικαίου, στους εισαγγελείς, στους δικαστές κτλ να τροφοδοτούν τις εργασίες τους σε καθημερινή βάση από την ευρωπαϊκή αυτή παραγωγή δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει και προσπάθεια σε ποσοτικό επίπεδο και έχουμε κάποια παραδείγματα με το 7 ετές πρόγραμμα όταν αναφέρεται σε δείκτες λέγει ότι ο αριθμός των περιπτώσεων δικαστικής διαμεθοριακής συνεργασίας είναι δείκτης θα έλεγα της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού νομικού συστήματος. Ο αριθμός των περιπτώσεων συνεργασίας. Αυτό είναι σημαντικό παράδειγμα, αλλά είναι λίγο γενικό λόγο όμως. Είναι θα έλεγα ένα μοναδικό παράδειγμα το οποίο δεν αρκεί από μόνο του. Πρέπει να γνωρίζουμε και γιατί σαν παράδειγμα ο αριθμός αυτός των περιπτώσεων συνεργασίας είναι τόσο χαμηλό σε σχέση με το σύνολο των υποθέσεων που θα μπορούσαν να καλυφθούν με τον τρόπο αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την πρακτική χρησιμότητα της προσφυγής στη δικαιοσύνη μέσω της αντίληψης που έχει ο Ευρωπαίος για την αποτελεσματικότητα των δικαστικών διαδικασιών. Μια αίσθηση δηλαδή την οποία πρέπει να έχει και όχι κάτι το οποίο ε, διαμορφώνει κανείς σαν αντίληψη μέσω μιας λεπτομερούς ε, ανάλυσης της κατάστασης. Η Επιτροπή με αυτά τα οποία προτείνει δείχνει αν θέλετε και την ε, πολύ μεγάλη αδυναμία του συστήματος οικονομικά. Κάτω του 1% 0, κάτι της 100 του προϋπολογισμού δεν υπολογίζουμε τα πάντα και την ποιότητά τους μέσω της δημοσιονομικής διαθεσιμότητας. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένας δείκτης ο οποίος λέγει ότι ο χώρος της Στοκόλμης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προτεραιότητα. Ενώ αντίθετα εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει. Η τρίτη γενική παρατήρηση είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι και αυτό όπως είπαμε τη σειρά του λίγο γενικόλογο. Η συγγήτρια έδωσε κάποιες αιτιολογίες σε σχέση με <clears throat> κάποιες λεπτομέρειες. Δεν έμεινε βέβαια στις λεπτομέρειες αυτές όσο θα έπρεπε και εγώ παρατηρώ ότι αυτό το γενικό λόγο της πρότασης επηρεάζει και όχι πάντα βέβαια θετικά πολλές από τις πλευρές από τις οποίες συντίθεται το πρόγραμμα αυτό. Κατανοώ βέβαια ότι οι στόχοι οι οποίοι περιγράφονται δεν είναι επακριβέστατοι, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί οι δράσης να μην είναι επακριβείς. Η, η μη επακριβής ακριβώς φύση των δράσεων αυτών στοιχειοθετεί σαφέστατα κινδύνους για την ίδια την ύπαρξη του προγράμματος. Σχετικά τώρα με το judicial training, την κατάρτιση των δικαστών κτλ. Και εδώ έχουμε προσπαθήσει σαν Επιτροπή Τζούρινγκ, νομική επιτροπή και θα το κάνουμε και στα πλαίσια της ΛΥΜΠΕ. Θα προωθήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση των δικαστών. Έχουμε κάνει κάποια βήματα. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις πρώτες ε, μετά από, τον, από τη συμφωνία της Στοκόλμης. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή της την προηγούμενη λέγει ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί σαφέστερα ο νέος δρόμος τον οποίο έχουμε σχεδιάσει στα πλαίσια της δικαστικής συνεργασίας. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα εδώ. Ο υπόλοιπο, ο άλλος πυλώνας αν θέλετε, ε, ε, του χώρου δικαστικής συνεργασίας είναι η συνεργασία σε επίπεδο αστικού δικαίου και σε επίπεδο ποινικού δικαίου. Και εδώ νομίζω ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να παρουσιάσει με πιο λεπτομερή τρόπο το πώς στηρίζει τη συνεργασία αυτή. Προφανώς και γίνονται κάποιες ποσοτικές αναλύσεις, προφανώς και γίνονται κάποιες ποιοτικές αξιολογήσεις. Το θέμα είναι με ποιο πρακτικό τρόπο θα ενισχύσουμε τους δικαστές των χωρών της Ένωσης έτσι ώστε να συνεργάζονται για να επιλύσουν τις τόσες πολλές διαμεθοριακές περιπτώσεις που χαρακτηρίζουν την δικαστική ζωή στην Ευρώπη τι υποστηρίζει εν πάση περιπτώσει, τι υποστηρίζει, τι δείχνει μάλλον η επιθυμία των δικαστών να συναντηθούν, να συνεργαστούν, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τις οποίες σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας. Λοιπόν θεωρώ ότι η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού έτσι όπως υποδεικνύεται, το monitoring, δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι αρκετά συχνό. Θα πρέπει να υπάρξει μια εποπτεία θα έλεγα πολύ πιο τακτική και πολύ πιο συχνή. Τελείωσα εδώ με την εξής παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει ένα ενιαίο πρόγραμμα που είναι το άθροισμα θα έλεγα των προηγουμένων προγραμμάτων της προηγούμενης προ... Ε, επταετίας, τις γνωστές αυτές πολιτικές στον τομέα της δικαιοσύνης. Εγώ ήμουνα μέλος της Επιτροπής ε, Πολιτισμού μέχρι πρόσφατα. Και η Επίτροπος για θέματα πολιτισμού παρουσίασε ένα ενιαίο πρόγραμμα το οποίο ενσωμάτωνε τα προγράμματα τα επιμέρους. Και η πρόταση της Επιτροπής μας ήταν αρνητική από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν ξέρω αν πρέπει κάτι να μάθουμε από εδώ. Ίσως τα πράγματα εδώ να είναι διαφορετικά. Αλλά υπάρχει παρόλα αυτά η ανησυχία να δημιουργηθούν συγχύσεις ανάμεσα στις διάφορες συνιστώσεις του προγράμματος. Σίγουρα στα πλαίσια του εξορθολογισμού θέλουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργώντας ορθολογικά να αποτρέπει επιπλέον και υπερβολικές δαπάνες, να επιτρέπει και σωστή και συγκεκριμένη χρήση των διαθεσίμων πιστώσεων. Λογικό αυτό. Παρόλα αυτά εδώ αναδύεται μία ανησυχία. Η δραστηριότητα του εκτελεστικού εδώ μήπως διαφεύγει μια αξιολόγηση και του δέοντος ελέγχου από πλευρά των κοινοβουλευτικών δομών έτσι ώστε όλες οι φωνές που ασχολούνται με το θέμα αυτό και όλες οι θέσεις του προϋπολογισμού που πρέπει να χρηματοδοτηθούν να διαφεύγουν κοινοβουλευτικού ελέγχου. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εδώ και με τις μετακινήσεις χρηματοδοτήσεων χωρίς έλεγχο από τη μία θέση στην άλλη, κάτι το οποίο μας δημιουργεί αμφιβολίες. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάναμε στην Επιτροπή Πολιτισμού, ότι εμείς θέλουμε να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα στις θέσεις αυτές. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε αμφιβολίες. τώρα παρακαλώ, εισήγησε την Επιτροπή μας ο Σύντομα, Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στην κυρία Μίχου για την ε, παρουσίαση του προγράμματος και τον εκπρόσωπο της Προεδρίας της Δανίας. Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη 2014-2020 έχει κατά εύστοχο τρόπο επιλέξει να συνδυάσει, να συνενώσει διάφορα προγράμματα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε προσφυρή εναρμόνιση. Ένα πολύ καλό δηλαδή σημείο κίνησης από πάσα περίπτωση. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες ερωτήσεις, σχόλια επίσης και να επισημάνω κάποια προβλήματα που απορρέουν από την πρόταση. Στο σύστημα που έχουμε τώρα διαπιστώνεται ανισορροπίας προς την γεωγραφική κατανομή των έργων και των προγραμμάτων. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Σε ποιο βαθμό θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να καταλήξει μια καλύτερη γεωγραφική διασπορά πλέον. Διότι οι ανισορροπίες πιστεύω σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στο γεγονός ότι οι διαδικασίες για όποιον θέλει να διεκδικήσει τέτοια ενίσχυση είναι πολύ περίπλοκες. Θα μπορούσαν λοιπόν να προστευτούν αυτές οι διαδικασίες. Και σημαντικό είναι πιστεύω να θεσπιστούν σαφή κριτήρια πράγμα το οποίο θα αποβεί οφέλο και τη Ένωση, βέβαια, αλλά και των πιθανών δικαιούχων και θα διευκολύνει, θα απλουστεύσει την πρόσβαση στο σύστημα. Ποιοι είναι οι στόχοι της Επιτροπής για τη γεωγραφική τουλάχιστον διασπορά των έργων. Άλλο πρόβλημα που έθιξε και ο κύριος Περλιγκέρ είναι ότι είναι κάπως ασαφής διατύπωση αρκετές διατάξεις όταν γίνεται λόγο για ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, Φρεφερρυπίν, που απαιτείται για να είναι δικαιούχος κανείς ε, ε, για βοήθεια. Ή αντίστοιχα, γενική, γενικόλογη διατύπωση των δικτών που επιτρέπει να διαπιστωθεί αν επιτυχάνονται στόχοι. Όλα αυτά είναι πολύ ασαφή η δε μεσοπρόθεσμη έκθεση που προβλέπεται για τα μέσα του 2018 νομίζω ότι θα έρθει, θα αργά. Γιατί ήδη θα πρέπει τότε να έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για την περίοδο μετά το 2020. Ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τη διαφάνεια, που επίσης θεωρώ πολύ σημαντική, θα πρέπει πιστεύω να προσπαθήσουμε να δημοσιεύσουμε έναν ε, κατάλογο δικαιούχων που επίσης δεν προβλέπεται τώρα στην πρόσταση της Επιτροπής. Γιατί δεν προβλέπεται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ε, γίνει η προσαρμογή, γιατί πολύ συνάρτηση στο Κοινοβούλιο βλέπουν ότι υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις και τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Σιγκλά. Ακούσαμε τον εισηγητή. Ας δούμε και τους συναδέλφους, τους λοιπούς συναδέλφους που ζητούν το λόγο. Κύριος Φάντεν Κάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ ολλανδικά. στον συγγνώμη, ξε... Ε, ξεκινώ ε, γιατί ήρθα με καθυστέρηση. Είχα 40 φοιτητέ που επισκέπτονταν και προφανώ δεν μπορούσα να του ε, αφήσω να περιμένουν, να του αγνοήσω. Η ομάδα του ΕΛΚ λοιπόν υποστηρίζει τι ευρείε γραμμέ τη προσέγγιση που μα παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημένοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε από κοινού στην ε, ε, απλούστευση και συγχώνευση των έργων ναι, για των προγραμμάτων ναι, αλλά χωρίς να χάσουμε και τις προτεραιότητές μας. Γιατί για μας κύριο πρόβλημα στην Ένωση είναι η κατανομή των κονδυλίων που έχει σαν αποτέλεσμα να παίρνει ο καθένας από λίγο κάτι για τη Στοκχόλμη, κάτι για την πρόληψη στα ναρκωτικά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, αλλά δεν πρέπει να ε, λησμονούμε ποτέ ότι αυτό το κάτι θα πρέπει να πηγαίνει στο καλύτερο δυνατό πρόγραμμα. Και πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, πιο θαραλέοι, να λαμβάνουμε αποφάσεις με περισσότερη παρησία. Διότι δεν αρκεί και δεν είναι απαραίτητα καλή ιδέα να δίνουμε στους πάντες από λίγο. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν επιτυγχάνεται με ποιο τρόπο. Οι στόχοι που έχουν οριστεί εξασφαλίζονται. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες ε, μετρήσεις, υπολογισμούς πιο επακριβείς ως προς τις ε, ευθύνες γιατί έχω να πω ότι έχω έναν ε, ασκούμενο εδώ που ε, με βοηθάει στην ε, δουλειά μου και διαπιστώνω ότι είναι πολύ περιορισμένη η ενημέρωση από τις επαφές που έχουμε των δικαστών, των εθνικών δικαστών που ασχολούνται ε, με θέματα ευρωπαϊκά. Πολύ λίγο γνωρίζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο οι δικαστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια ιδιαίτερη. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκάντ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε Σωστή του Δημοκράτες, έχουμε την υποφαινομένη ως ε, σκιώδη εισηγήτρια, λέει κυρία Γκέντς. Για να δούμε. Ε, τι, τι γίνεται με αυτή το λεγόμενο σενάριο Β, την επιλογή Β, να έχουμε δηλαδή δύο αντί για έξι προγράμματα. Άκουσα τους προλαλήσαντε. και εγώ Νομίζω ότι χρειάζεται να τα και κάπως τα πράγματα. Ίσως δύο προγράμματα σημαίνουν περισσότερη αποτελεσματικότητα, απλούστευση, αλλά ταυτόχρονα το θέμα είναι η διαφάνεια. Πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι και θα έχουμε ένα σωρό διαφορετικούς στόχους. Τι θα γίνεται από μια, τη μία χρονιά στην άλλη. Πώς θα εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα του ορισμού, του καθορισμού των ετησίων προγραμμάτων και των αφορά την οικονομία των κονδυλίων. Γιατί από αυτού συμφωνώ με αυτού οι οποίοι έλαβαν το λόγο προηγουμένω. Επίση, τι θα γίνει όσον αφορά την υποπτία, την αξιολόγηση. Θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, δείκτε. Δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις κάποιων μέτρων. Δεν λέω ότι είναι το πιο καυτό πράγμα στη ζωή των Ευρωπαίων, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδειχτεί ότι είναι αυτά τα προγράμματα χρήσιμα. Αυτά θα πρέπει να προσέξουμε επομένω, τη διαφάνεια πρώτον, δεύτερον το, το πρόγραμμα εργασία, το περιχαρακώσουμε, η κατανομή των πόρων, του στόχου, γεωγραφική κατανομή, γεωγραφική κάλυψη και την ε, ισορροπία όσον αφορά του επιμένου κριτήρια οι και να πιο, πιο, πιο συγκεκριμένοι σε όλα αυτά πριν προχωρήσουμε. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Κύριε Ρισμπέκ, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ναι. Και εγώ χαιρετίζω αυτή την πρόταση. Έτσι πρόκειται να εκλογικεύσουμε τα τρέχοντα, υπάρχοντα, ισχύοντα προγράμματα. Επίση, θα είναι τώρα πιο αποτελεσματικά τα καινούργια προγράμματα και έτσι θα σταματήσουμε την κατάτμιση των μέτρων ε, από την άλλη μεριά βέβαια όπως και άλλοι συνάδελφοι και εγώ θεωρώ ότι είναι αποκατευτικό το πόσο λίγο βοηθά η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προπολογισμού. Θα πρέπει επομένω να μην δίνουμε αυτή την λάθος εικόνα αδυναμίας της μπροστά στα προβλήματα των Ευρωπαίων. Επομένως, έτσι θα προχωρήσουμε και βέβαια η πρεκαδότηση αυτή δεν είναι και τόσο, τόσο, τόσο εντυπωσιακή. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να προστατοριστούμε προς ό,τι θεωρούμε προτεραιότητα. Και με αποφασιστικότητα να χρηματοδοτήσουμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε ε, όλοι μαζί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βεβαίω, έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία, τα στοιχεία που αφορούν το χρονοδιάγραμμα, όπω τα είπε η Κομισιόν, όπω τα είπε το Συμβούλιο και βέβαια να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όσο είναι πιο γρήγορα. Ίσως να κλείσει το θέμα φέτος κιόλα. Γιατί θα πρέπει να προσέξουμε και τη μεθοδολογία μας. Το είπαν αυτό και άλλοι προελίσσαντες. Ακόμα είναι αρκετά αόριστο το πρόγραμμα. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής μας είπε ότι θα τα λένε για να μπορέσει να, να, να δουλέψει η φαντασία μας και να μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Ωραία, οπότε ας δουλέψουμε και εμείς να συμπροτείνουμε κάποιες κατευθυντήριες. Να τα συμφωνήσουμε. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε για τι προτεραιότητε, όπω είπαν οι συνάδελφοι, και γι' αυτό και θεωρώ ότι η βασική προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε η κατάρτιση των δικαστικών να, να βοηθηθεί, γενικά το, το, προσωπικό ε, της δικαιοσύνης γιατί ε, αυτό το οποίο εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είναι δυνατόν αλλιώ να φτιάξουμε αυτόν τον ε, χώρο δικαιοσύνης. Πρέπει να εκπαιδευτούν οι εμπλεκόμενοι παράγοντες. Και να μην μείνει λοιπόν μια ιδέα και περιεχομένου αυτός ο χώρο η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Τώρα, για την προσβασιμότητα σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να οργανώσουμε κάποιες ηλεκτρονικές πύλες, να προβληθούν τα προγράμματα αυτά με τρόπο καινοτόμο. Ούτω ώστε να δούμε πώς είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν όλα όσα ε, σήμερα μας παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία, να προβληθούν περισσότερο επομένω αυτά τα προγράμματα να απλουστευθούν και να είναι πιο προσβάσιμα στους Ευρωπαίους. Τέλος, πάντα πολλές μεθοδολογίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιους ε, δείκτες για την χρηματοδότηση και θα πρέπει επίσης να δούμε εκ των υστέρων τι έγινε με την αξιολόγηση των τριών προγραμμάτων που παρήλθαν. Θα ανοίξουμε μια ματιά, θα δούμε έτσι το λέω και διπλωματικά, γιατί υπάρχουν κάποια μικρά κενά. Κάποια κράτη που δεν, δεν πήραν ποτέ χρηματοδότηση, κάποια δεν συνεργάστηκαν, άλλα δεν δοκίμασαν καν να χρηματοδοτηθούν, κάποιες χώρες δεν ε, αντιπροσωπεύονται καν. Παρά επομένω την, ε, το ευρύ πεδίο του προγραμμάτων. Επομένω και εδώ θα πρέπει να επιτελέσουμε σημαντικό έργο απλούστευση, προβολή και όλα αυτά με τον δεδομένο περιορισμένο προπολογισμό. Άρα πολλά θα πρέπει και εδώ να κάνουμε, ξεκινώντα ακριβώ με την περιχαράκωση των βασικών ορισμών ενιών. Αυτά από πλευρά ε, φίλων δημοκρατών. Σας ευχαριστώ τόσο κοινό χώρο δικαιοσύνη. Ναι, με ένα θεμητό ιδεολόγημα, λέει ο κύριο Μπρό. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Να περτανεύει δικαιοσύνη. Αυτό όμω δεν πάει να πει ότι θα πρέπει να έχουμε εναρμόνιση των δικαϊκών συστημάτων, των νομικών συστημάτων, του, του, του, του δικαίου. Γιατί ο καθένα με διαφορετικού διάβλου το πετυχαίνει. Επίση, η εναρμόνιση του δικαίου δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητη προπόθεση Δικαθέσει ε, για να δούμε τώρα ποιε χώρε στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, ποιε χώρε στην Ευρώπη τέλο πάντων. Υπάρχουν κάποιε χώρε που φυλακίζουν τον κόσμο για τι πολιτικέ πεπιθήσει, απαγορεύουν πολιτικά κόμματα, παρά το ότι ε, ε, προσπαθούν να πετύχουν του στόχου του ε, με ελληνικό τρόπο και απαγορεύονται επομένω διάφορε απόψει. Α πούμε, τι έγινε το 2015 στην Αρμενία, τι έγινε, τι έγινε, έχουμε κάποιε μη πολιτισμένε χώρε ε, αυτό έχει καμία σχέση με δικαιοσύνη, με την ιστορία να ασχοληθούν οι ιστορικοί. Οι πολιτικοί δεν μπορούν να επιβάλλουν τέτοιου είδου ε, απόψεις, δηλαδή ιστορικές. Αυτό είναι ολοκληρωτισμό. Τώρα, πριν κανένα αποπειραθεί να μπορέσει να, να, να, να καπελώσει 27-28 φορές, θα πρέπει, θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσει ότι αυτό το οποίο θέλει να επιβάλλει είναι σαν, σαν ιδέα δίκαιο. Και ότι η δική του χώρα είναι ίδια θα Έχουμε και, επίσης ε, και κάποια δικονομικά μέσα, ας πούμε το, το, ευρωπαϊκό ένταλμα, που αυτά δεν βοηθούν αντικειμενικά. Φυλακίζεται κόσμος, προφυλακίζεται χωρίς να έχουν γίνει, ε, οι, οι, να έχουν γίνει δίκες, ε, δεν τηρούνται αυτά τα οποία τα δικονομικά προαπαιτούμενα για την χώρα η οποία ε, εκδίδει, απελάβνει τον ε, φυλακιζόμενο. Οπότε προσοχή στο πώς χτίζεται έτσι τούβλο τούβλο του πετραδάκι πέτρα, στην Ευρώπη. Ναι, είναι αλήθεια ότι τα ψώνια είναι ευχάριστα. Shopping therapy, αλλά προσοχή δεν είναι δυνατόν κανένας να, να κατρακυλάσει κάποιες απόψεις για τόσο σημαντικά θέματα. Κύριε Μίχου θα θέλετε τώρα να λάβετε τη σκητάλη κατόπιν όλων αυτών τα οποία ακούσαμε και μετά να στραφούμε και πάλι στους ηγητές να ανθρολογήσουν για να κλείσουμε. Μίχου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μπορέσουμε να σας πούμε τις απόψεις και ο καθένας να πει στον άλλο τι θεωρεί, ε, τι πιστεύει για αυτές τις προτάσεις και οπότε και εγώ θα πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ μαζί σας σε ορισμένα θέματα 100%. Παρακαλώ επίσης συνεργαστείτε μαζί μας τους αμέσως επόμενους μήνες. Κάτι τώρα το οποίο όμως θα πρέπει να σας πω είναι το εξή. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και αν αυτή την προεκόντηση δεν είναι τόσο σημαντική, ε, ε, αυτό το, το όραμά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν επομένως σας δίνει την εντύπωση αν δίνετε κάποια ερμηνεία στα που είπα, ε, και, εγώ φταίω. Ακόμα και αν θεωρείτε ότι επομένω δεν πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μα δίνουν τώρα είναι περισσότερο από αυτό που μα δίνανε προηγουμένω. Γι' αυτό και εμεί θεωρούμε ότι είναι, είναι καλό ο προηγούμενο αυτό και θα πρέπει επίση γι' αυτό να τον εντοπίσουν, να τον ε, υλοποιήσουμε, να τον αξιοποιήσουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε του στόχου μα. Επίσης, άκουσα ένα σωρό παρατηρήσεις όσον την αυτών των προγραμμάτων. Μην ξεχνάτε. Επίσης, ούτε εμείς να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται να τρέξουν κάποια ετήσια προγράμματα εργασίας. Σύμφωνα με αυτά, κάθε δράση κατά λεπτός πρόκειται να καθορίζεται. Αυτό το οποίο τώρα έχουμε στα χέρια μας είναι ένα ευρύ πλαίσιο το οποίο αφορά τη μεθοδολογία. Πώς θα αξιολογούμε, ποιοι θα είναι οι δείκτες, τα κριτήρια. Άκουσα πάνω σε αυτό, ε, διάφοροι βουλευτές ε, είπαν ε, το, τα θέματα της, της αξιολόγησης, της, εποπτεία. εποπτείας. Όλα αυτά στου μέσου μήνε θα τα δούμε. Επίση, όσον αφορά την γεωγραφική κάλυψη, Οφείλω να σας πω επίσης ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια αυτά τα προγράμματα να, να, να διαδοθούν όσο γίνεται περισσότερο προς όλο τον κόσμο, προς τους ε, επιλέξιμους. Σύμφωνοι. Όμως δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κάποιους να ζητούν να γίνουν επιλέξιμοι. Άρα θα πρέπει εκεί να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας, ίσως να διευρύνουμε το πεδίο δράσης μας. Να κάνουμε περισσότερες, περισσότερες δράσεις και έτσι να μπορούμε να ελκύσουμε περισσότερο να συμμετάσχουμε από όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό σα λέω. Θεωρώ ότι αυτό που να κάνουμε και αυτό και θα κάνουμε και ξεκινάμε από αυτή τη χρονιά με τα σχετικά προγράμματα ε, με βάση τα όσα σήμερα ισχύουν. Επίσης, Έχουμε το τίσιο πρόγραμμα εργασία. Έχουμε το θέμα των, της υποβολής των εκθέσεων, τα οποία αποσκοπούν ή στο να υπάρχει διαφάνεια στην ανάλωση των χρημάτων προπολογισμού. Δεν το στρέψουμε εμείς. Εμείς θα είμαστε οι διαχειριστές αυτών των κονδυλίων. Και αυτό και για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η διαχείριση να γίνει με τρόπο που να εξυπηρετεί τους σκοπούς μας, αλλά να γίνει χρήστη, σωστή διαχείριση. Και σα ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Για να δούμε τώρα οι συγκεκριτέ μας τι έχουν να πει, να πούν για να κλείσουμε. Κύριε Κλάιτς, εσεί πρώτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι υπάρχει μια ευρυτάτη συνένεση πάνω σε ένα αριθμό αρχών στη διευκρίνηση ορισμένων στόχων που επιτρέπουν να προωθηθούν αρχές όπως η διαφάνεια. Περιμένω λοιπόν την επεξεργασία της έκθεσης αυτής σε συνεργασία με το Συμβούλιο, του εισηγητές και τον κύριο Μπερλίνγκουερ. Και εγώ θα είμαι τηλεγραφικός. Είναι αλήθεια ότι στα πλαίσια της συζήτησης μου φάνηκε ότι αναφαίνεται μια κάποια συνένεση. Θέλω να διαβεβαιώσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εμείς θα συνεργαστούμε στενά μαζί της. Αυτό έχουμε κάνει και μέχρι τώρα. και θα επιμείνουμε στις παρατηρήσεις μας έτσι ώστε να δούμε εάν η τελική έκθεση μπορεί να φανεί να λειτουργήσει θετικά στην προσπάθεια την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα δύο σημεία όμως να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω. Πρώτον, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συνεχή προσπάθεια σύγκρισης αυτού το οποίο γράφεται στους νόμους και στους κανονισμούς και αυτού το οποίο συμβαίνει καθημερινά στη ζωή του πολίτη. Είπαμε, η αρχή της implementation, λέει αγγλικά ο κύριος Μπερλίνγκουερ. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε οι πραγματικές συνέπειες των ρυθμίσεων αυτών να αφορούν τον πολίτη, να αφορούν την καθημερινότητά του. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τυπικό πρόβλημα ενός επταετούς προγράμματος, ίσως όχι ενός μόνο ετούς. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις της τεκμηριωμένες των πολιτών. Τώρα σχετικά τα προγράμματα τα διετή και για την κατάρτιση των δικαστικών κτλ. Αυτά τα οποία ήδη κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Κοινοβούλιο θα πρέπει να οριστούν σωστότερα στα πλαίσια του επταετούς προγράμματος. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος όλους για τη συζήτηση η οποία προηγήθηκε. Να ευχαριστήσω τα μέλη, τα εκλεκτά της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που πήραν μέρος στην κοινή συζήτηση. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπερλίνγκουερ, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα τώρα. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον εκλεκτό συνάδελφο. What is this? Yeah, the program, establishing Ah, yes, yes, yes, yes, yes. I jumped over the point number 17. Έχασα το σημείο 17. Το σημείο 17 αφορά την κατάρτιση του προγράμματος Δικαιώματα και ηθαγένεια. Έχουμε ανάμεσά μας την κυρία Κίνγκα Γκένς. Αλλά και εδώ υπάρχει παρουσίαση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Παρασκευή Μίχου πάλι θα μας παρουσιάσει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για δράσεις με προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία στα πλαίσια της δημιουργίας ενός χώρου στον οποίο τα δικαιώματα του πολίτη θα είναι ε, θεμελιωμένα και θα πρέπει να προστατευθούν ακόμα περισσότερο. Αυτό το πρόγραμμα διαδέχεται τρία ισχύοντα αυτή την εποχή προγράμματας Πρώτον, θεμελιώδη δικαιώματα και ηθαγένεια, το δάφνη 3 και τρίτον, το τμήμα που αφορά την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων ενός ευρύτερου προγράμματος. Τα τρία αυτά προγράμματα λοιπόν συνενούνται για λόγους απλοποίησης και εξορθολογισμού, γιατί ο τομέας του δικαίου ε, μερικές φορές υποδεικνύεται σαν παράδειγμα πολυδιάσπασης. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στην κυρία Μίχου και μετά στον εκπρόσωπο της Προεδρίας. Θα ακολουθήσουν τα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να πάρουν μέρος στη συζήτηση. Κυρία Μίχου, ευχαριστώ για μια ακόμη φορά Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφραστώ για το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια Ίσως κάποια από αυτά τα οποία θα πω να θεωρηθούν επικάλυψη. Βλέπω ότι το ακροατήριο είναι το ίδιο, θα προσπαθήσω να αποφύγω τις επικαλύψεις και είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Ήδη στις 15 Νοεμβρίου παρουσιάσαμε το δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια για το 2014 μέχρι το 2020. Το τα υπόλοιπα προγράμματα για τη δικαιοσύνη σας παρουσίασα λίγο πριν. Προσπαθούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε το μέγιστο αριθμό συνεργειών και παρομοίων διαδικασιών έτσι ώστε να απλοποιήσουμε την κατάσταση και να διασφαλίσουμε μεταξύ των προγραμμάτων αυτών μεγαλύτερη κοινότητα. Η Επιτροπή προτείνει ένα δημοσιονομικό φάκελο ο οποίος φτάνει τα 449 εκατομμύρια κατέτος και έχει σαν στόχο να υποστηρίξει νομιθετικές και πολιτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσει επίσης τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την επιτυχή προσπάθεια την οποία ακολούθησαν μέχρι τώρα, η οποία έγινε μέχρι τώρα από τρία διαφορετικά προγράμματα. Το πρόγραμμα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια, το πρόγραμμα Δράφνη και το πρόγραμμα Progress, δηλαδή καταπολέμηση διακρίσεων και ισότητα των φύλων. Η συγχώνευση των τριών αυτών προγραμμάτων έχει σαν στόχο τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των δραστηριοτήτων χρηματοδότησής τους. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι εμείς δίνουμε λιγότερη σημασία σε ένα από οποιοδήποτε από τα τρία αυτά προγράμματα και στη χρηματοδότησή τους. Η αλλαγή της δομής του προγράμματος δεν σημαίνει ότι οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες των τριών προαναφερθέντων προγραμμάτων θα πάψουν να υπάρχουν. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαν στόχο να διατηρήσει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και να τις βελτιώσει αναπτύσσοντας περαιτέρω τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων. Ειδικότερα τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε θετικά την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα επιτεύγματα μέσω του προγράμματος Δάφνη. Υπογραμμίζει την σημασία την οποία θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον του προγράμματος Δάφνη, κάτι το οποίο υποστηρίχθηκε ε, συστηματικά από την εποχή της γέννησής του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αλήθεια ότι το όνομα Δάφνη δεν περιλαμβάνεται στον τίτλο του προγράμματος. Παρ' όλα αυτά, οι δραστηριότητες του προγράμματος Δάφνη καλύπτονται πλήρως στα πλαίσια της εμβέλειας του προγράμματος. Στα πλαίσια του νέου προγράμματος Δικαιώματα και Ιθαγένεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναπτύξει τις βέλτιστες δυνατές πρακτικές καταπολέμησης της βίας, ισότητα φύλων, και ανατροφής των παιδιών και δικαιωμάτων συγγνώμη των παιδιών που καλύπτονται από επιμέρους προγράμματα μέχρι σήμερα. Συνολικά το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια θα συνεισφέρει στην δημιουργία ενός χώρου στα πλαίσια του οποίου τα δικαιώματα των προσώπων θεμελιώνονται στη συνθήκη και στην χάρτα των ανθρωπίνων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο χώρος αυτός θα επιτρέψει να υπάρξει ουσιαστική στήριξη στις πολιτικές που προωθούν την ισότητα και καταπολεμούν κάθε μορφές διάκρισης. Θα διατηρήσει δραστηριότητες για επιμέρους, ε, χρηματοδοτήσεις για επιμέρους δραστηριότητες, θα αποτρέψει τη βία και θα προστατεύσει τα θύματα της. Θα συνεχίσει να πολεμά για τη συμπερίληψη και όχι αποκλεισμό των Ρωμά και η κοινωνία των πολιτών είναι κομβικός παίκτη για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Και γι' αυτό για όλες αυτές τις δράσεις θα συνεχίσουμε τη χρηματοδότησή τους. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει επίσης τα δικαιώματα των παιδιών, θα παράσχει τα απαιτούμενα δημοσιονομικά μέσα για την κάλυψη πρωτοβουλειών, όπως ε, η γραμμή 116.000 ε, αναφορά άσκησης βίας και κακομεταχείρισης παιδιών και άλλα συστήματα προειδοποίησης για την κακομεταχείριση των παιδιών σύμφωνα ακριβώς με τους τομείς τους οποίους τα παιδιά είναι σε κίνδυνο. Παράλληλα θα στηρίξει πρακτικά τις χώρες μέλη για την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πακέτου για την προστασία των δεδομένων που είναι σε φάση διαπραγμάτευσης και θα παράσχει ε, πιστώσεις για τη βελτίωση του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών. Να αναφερθώ ίσως πιο συγκεκριμένα σε κάποια από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Θα ήθελα να δούμε με διαφορετικό τρόπο τα προγράμματα αυτά όπως το κάναμε και στα πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος δικαιοσύνη που σας παρουσίασα. Στόχος μας πάντα παραμένει η ευθυγράμμιση, η απλούστευση και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Και η ευελιξία. Ευελιξία γιατί πρέπει να προσαρμόσουμε το 2014 έως το 2020 και να και για να ολοκληρώσω θα ήθελα να πω ότι και εδώ έχουμε αρχίσει συζητήσει με το Συμβούλιο και προσβλέπουμε σε συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ολοκληρώσουμε και αυτό το κομμάτι των προτασών μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Δηλίντε από το Συμβούλιο σας παρακαλώ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, μπορώ να είμαι πολύ σύντομο πέρα, ότι καλύφθηκαν οι παρατηρήσει μου στο μεγαλύτερο του σταθμό από την προηγούμενη μου παρουσίαση για το άλλο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, όπω είπατε, καλύπτεται από την ομάδα εργασία ad που παρακολουθεί παράλληλα τις προτάσεις. Μια λύση ορθολογική διότι προκύπτουν αντίστοιχα ζητήματα στι διαπραγματεύσει των δύο παράλληλων προτάσεων. Και όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε πίεση χρόνου όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό. Οι διαπραγματεύσει μέχρι τώρα δείχνουν γενικότερη υποστήριξη στην ομάδα εργασία από πλευρά των κρατών μελών για τη γραμμή που έχει οθετήσει η Επιτροπή για την αποσυντευξη και τον ε, εξορθολογισμό στην υπόθεση αυτή. Και περιμένω να ακούσω τι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και να αρχίσουμε και τι συζητήσει στο χειρότερο δυνατό με το Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σα ακούσουμε τώρα του βουλευτέ μα, Κύριε Μπουζούτσιλ. Α, η κυρία Κόλτς, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, η πρώτα. Είναι δύσκολο βέβαια να μιλήσω για το πρόγραμμα αυτό χωρίς να κάνω αναφορά και στο άλλο, αφού είναι αριλένδετα, το είπαν όλοι. Από την άλλη δεν θέλω και να επισέλθω σε λεπτομέρειες ε, ως προς τη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, γεωγραφική διασπορά που πάλι είναι κοινό στοιχείο με το άλλο πρόγραμμα. Θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό το εμπλακή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκαίρως ε, στον προγραμματισμό, στο ετήσιο πρόγραμμα. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε την, ε, μπορούμε να προβλέψουμε τι είδος προτεραιότητας θα έχουμε για το 2020, αλλά είναι πάντα πολύ σημαντικό να γίνει προσεκτικά η προετοιμασία και να έχουμε αποτελεσματική χρηματοδότηση και χρήσιμη. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής μίλησε και εκείνη για αποτελεσματικότητα, πλούστευση. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Απλούστευση που έχει σημασία σε δύο πράγματα. Στη διαχείριση βέβαια των λογαριασμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πολύ σημαντικό είναι να προσταθούν και οι κανόνε λειτουργία και η διαχείριση των ε, ταμείων για τον κάθε ένα δικαιούχο που θα απευθυνθεί στα ταμεία αυτά, γιατί υποφέρει πολύ ο κόσμος. Ας προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων. Ένα κομμάτι που αφορά περισσότερο την πτυχή της Ιθαγένας είναι πιο συγκεκριμένο και νομίζω ότι μπορούμε να προβλέψουμε το τι πρόκειται να συμβεί και να ορίσουμε προτεραιότητα. Τα άλλα κομμάτια όμως είναι λιγότερο συγκεκριμένα. Και εν προκειμένου θα ήταν σημαντικό να μας απασχολήσει το μέλημα της ευαισθητοποίησης γιατί είναι λίγοι τελικά οι πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν τι συνέπειες για τα δικαιώματά τους έχει η συνθήκη της Λισαβόνας, σε ποιο βαθμό μπορούν να στηριχθούν σε αυτήν. Και το έχω επισημάνει ότι χρειάζεται περαιτέρω ε, δουλειά στον τομέα αυτών. Γενικά πρέπει να ενισχυθούν ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά πολέμηση των ε, διακρίσεων, των ξενοφοβικών συμπεριφορών και που βλέπουμε άλλωστε ότι εντείνονται στην Ευρώπη και ίσως να είναι πολλοί οι πολίτες οι οποίοι αισθάνονται να μην ε, διαφυλάσσονται, να μην, να μην προστατεύονται τα δικαιώματά τους. Ε, αναφέρατε και εσείς τους ομοφυλόφιλους παρενδυτικούς και άλλους που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και που θα πρέπει να διαφυλάξουμε. Επίσης, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και ε, κίνητρα για την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων. Μιλώντας δε για τα δικαιώματα των πολιτών, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι απαραίτητο να διαφυλαχθούν οι αρχές της Ένωσης, θεμελιώδη δικαιώματα, δημοκρατία κτλ. που ουσιαστικά αποτελούν την εγγύηση για τα δικαιώματα των πολιτών. Παιδιά, όταν πηγαίνουν στο σχολείο δεν επιτρέπεται να ε, μην ενημερώνονται πλέον. Πρέπει να υπάρχει η ευαισθητοποίηση η οποία θα αλλάξει μακροπρόθεσμα τις νοοτροπίες. Χρειάζονται λοιπόν ειδικά προγράμματα με εμπλοκή του και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πρόγραμμα εργασίας και στα διάφορα, στον προγραμματισμό για τα διάφορα έτη και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον η Επιτροπή μας δεν θα μπορέσει να έχει τις αποφάσεις για τα χρήματα, για τα κονδύλια. Αυτό είναι αρμοδιότητα άλλων αλλά μπορούμε να συζητήσουμε τον προγραμματισμό τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κότς. Κύριος Μπουσούτηλ. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριος Μπουσούτηλ. Εγώ λαμβάνω τον λόγο για λογαριασμό της κυρίας Αντζελίλη, της κοιόδου εισηγητρίας του ΕΛΚ, διότι σήμερα έπρεπε να συναντήσει, μάλλον μαζί με τον ε, πρόεδρο Σούλτ να μιλήσουν στην Ελληνική Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ε, σήμερα. Εμείς πάντως οπωσδήποτε μπορούμε παρά να χαιρετίζουμε το γεγονός ότι με αυτή την πρόταση εκλογικεύεται, απλουστεύεται η κατάσταση, ε, μια που έχουμε αυτή την συνένωση προγραμμάτων πρωτοβουλειών, σε μια ενιαία δεσμή μέτρων. Βεβαίω και αυτό την μπορεί παρά να μα βρίσκει σύμφωνο. Διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να σταματήσει η διασπάθηση των πόρων και ε, περιττή γραφειοκρατία και διοικητικές ενέργειες που τώρα είναι δυνατόν επομένως να διοχετεύονται να ξεκινήσουμε αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με κάποια επιμέρους στοιχεία στην πρόταση, κάποια στοιχεία τα οποία για μας έχουν σημασία. Ας πούμε, η γενική στόχη, ο γενικός στόχος του προγράμματος Θέλουμε να καλυφθούν και τα δικαιώματα των ανηλίκων. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Η αναγνώριση της σημασίας της επίτευξης των σκοπών του προγράμματος μέσω κατάρτισης και συνειδητοποίησης. Επίσης και με κάποιους είναι σχετικά υποστηρικτικά δίκτυα. Επίσης η φιλοδοξία του να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες χρηματοδότησης με κάποιο είδους προσέγγιση με μεγαλύτερο προσανατολισμό, εστιασμό ή στα αποτελέσματα. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η πιο δόκιμη ε, μεθοδολογία. Επίσης, να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά την συμπερίληψη ή στις δράσεις του προγράμματος το πώς θα βοηθηθούν ε, κάποιο είδους ε, βασικά ευρωπαϊκά δίκτυα που συνδέονται με τους σκοπούς του εν λόγω προγράμματος. Η κυρία Αντζελίλη επίσης μου είπε να σας διαβιβάσω ότι Έχουμε μια σειρά μη κυβερνητικών οργανώσεων που ήδη έχουν τις επαφή μαζί τη και έχουν προτάσεις και θέλουν μέσω τροπολογιών αυτές να προωθηθούν εις το συζήτησή μας. Και έχουμε τον λόγο κονδύλιο το οποίο προαναφέρθηκε το 116.000 και αφορά αυτό το στο δίκτυο, αφορά επίση αυτό το, την, τον ενιαίο του τηλεφωνικό αριθμό. Τέλος πάντων, αυτό το κονδύλιο το οποίο πρόκειται να ε, βοηθήσει όλους τους επιλέξιμους του προγράμματος. Αυτά όσον αφορά το ΕΛΚ. Πάντως, πρόκειται εν καιρό να σας υποβάλουμε και πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει η κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστούμε και εμεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την παρουσίαση. Νομίζω ότι οι στόχοι που ετέθησαν είναι πάρα πολύ θεμητή, επενετή, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα όσα σήμερα ισχύουν για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τι θα γίνει με πολίτε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τι δυσμενεί διακρίσει, την ε, ισότητα και, τα θέματα γεωνική αλληλεγγύη. Τώρα για να ε, να προσθέσουμε τη διαδικασία, θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε όντως μια προσέγγιση ε, μια προσέγγιση η οποία να έχει σχέση με τα αποτελέσματα, οπότε χρειάζεται εδώ πέρα ε, να πρετανεύσει η συνέργεια, να είμαστε αποτελεσματικοί. Ε, Βεβαίω θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε εδώ και κάποια, α, κάποιες λεπτομέρειες που έχουν σημασία, αλλά εδώ έχουν ε, έχουν παραλυφθεί γιατί ακριβώ ο διάβολο κρύβεται στη λεπτομέρεια. Ε, τι να κάνουμε, ισχύει αυτό. Επομένω. From the Commission, how they plan to proceed to conduct a strategic work on violence. Να συνεχίσουμε να καλύπτουμε και με αυτό το πρόγραμμα, όπως και με το Δάφνη και με το Δάφνη 3 να καλύπτουμε τα θέματα της βίας κατά και γυναικών. προσοχή γιατί αυτό μας παρακολουθεί πάρα πολύ το ότι όταν γίνει αυτή η προγραμμάτων δεν θα καλύπτονται αρκετά τα θέματα τη ισότητα. θα εκτιμούσαν πάρα πολύ να μας διασκεδάσει τις εμβολίες μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω και κάποια άλλα πράγματα που με προβληματίζουν αυτά τα οποία αφορούν το άρθρο 4. Το, η δεύτερη παραγραφός εδώ αναφέρει ένα σωρό θέματα, ε, ένα σωρό στόχους. Προσοχή, μην ε, σκιάσει μία την άλλη. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει σαφήνεια, να είμαστε σίγουροι ότι ο κάθε σκοπός του προγράμματος έχει την προσοχή που αρμόζει. Επίσης να αναφέρουμε και την ξενοφοβία, να αναφέρουμε τις, ε, τον εξτρεμισμό, γιατί με, με την, ξεν, με την ξεν, ξενοφοβία και τον ε, εξτρεμισμό έχουμε φαινόμενα τα οποία ολοένα και επεκτείνονται. Άρα θα πρέπει να υπάρχει καταπολέμησή τους και θεωρούμε ότι δόκιμος τρόπος είναι αυτά τα προγράμματα. Γενικά πρέπει να σας πω ότι με προβληματίζει το κατά πόσον ε, η ισότητα των φύλων ε, καλύπτεται ακριβώς όπως και δυσμενείς διακρίσεις ε, και κυρίως διακρίσεις κατά των ε, ατόμων με δικές ανάγκες. Θα πρέπει αυτά με πιο συγκεκριμένο τρόπο να καλυφθούν, να μνημονευθούν Αυτές είναι οι βασικές μου αρχικές παρατηρήσεις κύριε Πρόεδρε και περιμένω πώς και πώ το να συνεργαστούμε στα πλαίσια ε, αυτού του νομοθετήματος και με την κυρία Γκάινς και με τους άλλους ε, σκιώδεις εισηγητάς, αλλά να συνεργαστούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ευχαριστούμε, εμεί ευχαριστούμε, λέει ο κύριο Λόπε Αγγελάρ και δίνει το λόγο στον κύριο Κέρκχομπ. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι να σα πω σε αυτό το στάδιο. Όμω, όμω, όμω να σα τονίσω ότι θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις φιλοδοξίες που έχουμε. Αυτό ισχύει για κάθε πρόγραμμα. Αυτό είναι θεμητό, αλλά κανείς θα πρέπει να προσέχει. Να προσέξει. Πού θα εστιάσει την προσοχή του. Ο καθένα, έχει ένα σωρό επιθυμίες. Όμως όσο πιο πολλέ επιθυμίες πιο δύσκολο είναι να καλυφθούν. Και αυτό τελικά καταλήγει σε ματέωση, σε απογοήτευση. Έχουμε τώρα το θέμα της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της συνειδητοποίησης σε σχέση με το τι μέτρα λαμβάνονται για τους Ευρωπαίους, για τους νέους. Πού μπορεί να ταυτιστεί λοιπόν ο, ο νέος με αυτά τα προγράμματα, Πώς μπορούν να βοηθούν οι σχέσεις μεταξύ των νέων στις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Ό,τι προβλέπει αυτά τα προγράμματα να το μεταρρυθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και έχουμε και αυτά τα κέντρα πληροφόρησης, όπως έχει εδώ και το Κοινοβούλιο. Και, εάν κανείς έχει το σωστό μήνυμα και το προθεί με το σωστό τρόπο, τότε αυτό αποδίδει. Πολλές φορές. Ε, οι νέοι δεν ξέρουν τι προβλέπεται, έστω και αν είναι προς όφελος τους. Άρα, προσοχή. Να ξέρει κανείς τι υπάρχει, τι διατίθεται. Άρα να ξέρουμε εμείς ότι θα υπάρχει σωστή, αποτελεσματική ενημέρωση. Γι' αυτό και έχει το κοινοβούλιο αυτά τα γραφεία παντού στον κόσμο. Όσον αφορά την παιδεία και την εκπαίδευση, Αναμφίβολο. θα πρέπει να συνεχιστούν οι πρωτοβουλίε μα. Τελικά, η... Ναι. Πολλέ φορές μένουν στο περιθώριο των πολιτικών μας. Εγώ με τα διαθέματα που τους καίνε και τα οποία έχουν να κάνουν άμεσα με την Ευρώπη. Για κολλήνω.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 E και επίσης θέλουμε να έχουμε ένα γιούρας ε, καλύτερο όσον αφορά την κινητικότητα και επίσης να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Επίσης, ε, αυτό το οποίο εδώ θέλουμε είναι να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά κάποιες ε, διαδικασίε, διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης γιατί ο κόσμος θέλει να ξέρει περισσότερα για αυτό το, το, το portal e Justice ή το Justice Online και επίσης να υπάρχει αυτή η ενημέρωση που να καλύπτει όλα τα κρατημέλη. Το, το σπουδαίο είναι ότι στα πλαίσια αυτής της ε, έκθεσης να τονώσουμε τον προβληματισμό, τον προβληματισμό όσον αφορά τις επιπτώσεις ε, αυτών όλων, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους. Θέλουμε συμμετοχική δημοκρατία και επίσης πρέπει οι Ευρωπαίοι να μπορούν να έχουν ε, μια ενημέρωση για όλε τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Κοινοβουλίου. Τώρα, ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να προβούμε σε κάποιον συνδυασμό, και περιμένουμε πώ και πώ να ακούσουμε τι έχει να προτείνει το Συμβουλίο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι ε, στην τελευταία μα συνεδρίαση δεν μπορέσαμε να ακούσουμε αυτά τα οποία είχαν προτείνει αυτά τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ κύριε Βοδοπούλου και ο κύριο Λόπε Αγγελάρ και πάμε τώρα παρακάτω όπου θα πρέπει να ακούσουμε τι έχει να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θέλετε το λόγο, μάλιστα. Έχετε το λόγο, κυρία. Ευχαριστώ που δίνετε το λόγο. Κύριε πρόσωπο Επιτροπή. Ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο και όλες τις επιτροπέ Επιτροπές για τις εντροπολογίες τους. Νομίζω ότι έτσι πρόκειται να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, ε, η συμμετοχή, η δυναμική των ε, Ευρωπαίων. Τώρα, ή στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής κρίσης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτες να είναι κοντά στην καρδιά, στο επίκεντρο της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια από αυτή τη δράση αποσκοπεί να κάνει την ζωή τους πιο εύκολη. Άρα και εμείς θέλουμε να υπάρχει μια τέτοια επαφή με τους ε, πολίτες. Να μιλάμε για τον άνθρωπο, όχι για τις αρχές και τις θεωρίες. Να, λοιπόν, ποιε αρχέ διαπνέουν τι προτάσει μα. Τώρα, όσον αφορά την νομική φάση. Αντιλαμβανόμεθα τι θέλει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, γιατί θέλετε να αναφερθούν ρητό όλε οι μέρου αρχέ που διέπουν την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Εκλέγει, εκλέγεστε, του την προ το κοινοβούλιο, το ξαναφέρνει στο κοινοβούλιο κλπ. Όλα αυτά όμω. Να κάνουμε το άρθρο 20 για τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λέει αυτά και το πρώτο άρθρο τη πρότασή μα, το οποίο νομίζω ότι καλύπτει αυτά τα δικαιώματα. Και οπωσδήποτε αυτό το οποίο εμεί θέλουμε είναι, είναι να, να, να ενημερώνονται οι πολίτε για όλα τα προαναφερθέντα. Επίση, ε, θέλουμε με, να γίνεται μια δημόσια διαβούλευση και εμείς προτείνουμε δύο συναντήσεις στα κρατημέλη. Στα γραφεία της Επιτροπής. Έχουμε, έχουμε, υπάρχει διάλογος με την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς της. Τώρα σαν αφορά τον προπολογισμό. Όντως, περιορισμένη είναι η χρηματοδότηση. Για ποιο λόγο. Πρώτον, τόσο επιτρέπει, αυτά τα περιθώρια μας δίνει, στους και κεφάλαιο του προπολογισμού. Δεύτερον, θεωρούμε ότι μια είμαστε σε εποχές δεν είναι σωστό να εκταμιεύουμε μεγάλα ποσά ε, για δραστηριότητε επικοινωνία. Τρίτον, το θέμα δεν είναι μόνο ο προπολογισμό. Είναι το πώ θα έχουμε συνέργεια. Γι' αυτό και θέλουμε να κινητοποιήσουμε τα θεσμικά όργανα, όλους. Επομένως, οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να βοηθήσουν με κάποιες συμπληρωματικές δραστηριότητε μέσα των ίδιων πόρων. Ήδη έχουμε αρχίσει αυτή τη διαδικασία. Με δεδομένο λοιπόν το χρονικό πλαίσιο που έχουμε για να ενεργήσουμε, να προχωρήσουμε ευθύ αμέσω ή στην πρώτη ανάγνωση ή στι προπαρασκευαστικές κινήσεις πλήρη συνεργασία με όλα τα θεσμικά και ιδίω με το Κοινοβούλιο. Επίση. Είπατε ότι θέλετε να παραέχουμε πολλούς στόχους. Αυτό που μπορεί να γίνει μέσω κάποιων φορέων να ακούγεται η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών. Επομένως, με την έκθεση για, για τους Ευρωπαίους θα ρυθμίσουμε πολλά θέματα εφαρμογής νομίζω ότι θα μας βοηθήσει το να συμφωνήσουμε, το να τα βρούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και άρα θα καλύψουμε και τις προσδοκίες των πολιτών. Ευχαριστούμε. κύριο Λίν, για το Συμβούλιο. Από πλευρά του Συμβουλίου εγώ έχω να σας πω ότι θεωρούμε πάρα πολύ θετικό είναι το σχέδιο κειμένο του εισηγητού. Επίσης, θεωρούμε ότι επίση ε, έχουν ληφθεί υπόψη διάφορε τροπολογίε βουλευτών. Και το Συμβούλιο μπορεί τώρα να ξεκινήσει την εξέταση του σχεδίου εκθέσεως και τις λοιπές τροπολογίες. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο μετά από προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν, ε, έγιναν δεκτές θετικά θα έλεγα και έχουν υπάρξει ελάσσονος στο οικολογίες. Δηλαδή το Συμβουλίο υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να υπάρξει ένα συγκεκριμένο στόχος για το έτος του πολίτη το 2013. Η πρόταση παρατηρεί με πολύ ενδιαφέρον ακριβώς τους στόχους και της Επιτροπής σας. Ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα διάφορα θέματα στο σωστό τους πλαίσιο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το χρονικό πλαίσιο και το οικονομικό πλαίσιο. Και γι' αυτό πρέπει να ορίσουμε σωστά τους στόχους μας το 2013. Για το 2013. Θα εξετάσουμε την πρόταση θεωρώντας ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε να ξεκινήσει τις προετοιμασίες η Επιτροπή. Αν δεν πάρουμε γρήγορα απόφαση φοβάμαι ότι θα δυσκολέψουμε τα πράγματα και σε επίπεδο προετοιμασίας. Η πρόταση εδώ Νομίζω είναι μια καλή πρώτη βάση συζήτησης και μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να πάρουν τα μέτρα που απαιτούνται έτσι ώστε η πρωτοβουλία αυτή να εξελιχθεί θετικά. Ευχαριστώ πολύ τώρα. Θα ακούσουμε τους ε, συναδέλφους. Κύριε Γκρίσπεκ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ την Αντιγόνη Παπαδοπούλου για την έκθεση, για τα σχόλια. Οι τροπολογίες μα ήρθαν μόλις σήμερα και μόνο στα αγγλικά δεν είχα το χρόνο να τις εξετάσω στις λεπτομέρειές τους. Πάντως είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την από το ενδιαφέρον την επιλογή των συναδέλφων 114 τροπολογίες και πάντως αυτό αποτελεί εκ μέρους των βουλευτών αναγνώριση και δείγμα της σημασίας που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια το έτος του Ευρωπαίου πολίτη. Η ηθαγένεια πιστεύω θα πρέπει να καταστεί κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι χωρίς Ευρωπαίο πολίτη Ευρώπη δεν υπάρχει. Ευρώπη δεν μπορούμε να χτίσουμε και κυρίως μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης που γνωρίζουμε, αλλά και κρίσης αξιών που γνωρίζουμε και έτσι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Άκουσα του εκπροσώπου και τη Επιτροπή και του Συμβουλίου και έχω την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι συνενετικό και αυτό ω προ τι ε, θέσει του, στι θέσει που ακούστηκαν σήμερα, που ε, κάνει μια προσπάθεια να ανέβει, να κατέβει μάλλον ε, μια κυλιόμενη σκάλα που όμως πάει προς τα πάνω το, η εικόνα δεν ξέρω αν είναι σαφής, αλλά πάντως την ώρα που προσπαθούμε, που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αδιαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αποξένωσης που αισθάνεται ο πολίτης εναντί αυτού του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή την ισχνή αίσθηση ε, του ανήκειν σε αυτό το οικοδόμημα, δίνουμε πολύ περιορισμένα μέσα και προβλέπουμε δράσεις που υπολείπονται πολύ των στόχων μας και των ανακών μας. Ε, ευχαριστώ λοιπόν και εγώ. Έχω καταθέσει δικέ μου τροπολογίες οι οποίες ιδιαίτερα με ενδιαφέρουν. Για να εξηγήσω πολύ γρήγορα, η πρώτη μου τροπολογία ε, στόχο έχει να διευρυνθεί το 2013 όχι μόνο στην ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και να καλύψει ε, η θεματολογία του έτους κάθε πτυχή της ε, ε, ζωής, βιώσιμη ανάπτυξη, κατάρτιση, ισότιμη μεταχείριση, όλα αυτά τα οποία αποτελούν δείκτες και στοιχεία του ανήκειν στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Επίσης ιδιαίτερα από τις, με τις τροπολογίες θέλω να επιμείνω στα ζητήματα της ε, δικαιοσύνης, μια και εμείς στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών ίσως αυτό να οφείλεται στην ε, τη της να με αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ο χώρος της δικαιοσύνη ελευθερίας και τη ασφάλεια πρέπει να μην χάνεται από τις προτάσεις και βλέπω ότι αναφέρονται συχνά οι επιβάτες, τουρίστες και τα λοιπά στο κείμενο, αλλά όχι οι ελευθερίες. Δεδομένου ότι πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε τους πολίτες για τη χρονιά αυτή, ε, για τα δικαιώματά τους, πρόγραμμα της Στοκχόλμης πάνω απ' όλα, καταθέτω τις τροπολογίες μου με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το χώρο της δικαιοσύνης τον οποίο τόσο συχνά συζητούμε, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δικαίωμα στην ενημέρωση και όλα τα θεμελιώδη ε, κείμενα τα οποία μας απασχολούν στις εργασίες μας. Επίσης, οι διαδικτυακές πύλες με ενδιαφέρουν ιδιαίτερο, το EURES, το Injustice, αποτελούν ε, στόχο, πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους και η ορατότητα αυτών των πυλών και η πρόσβασιμότητα για τον κάθε πολίτη. Ιδιαίτερα θα ήθελα να υπογραμμίσω μία πτυχή, το, την αρχή της πολυγλωσίας. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δούμε πώς οι, οι δράσεις μας και οι προσδοκίε μας να προβάλλονται να είναι ορατές από όλους. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα το καταφέρουμε όλο αυτό ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ε, φέτος, ε, να δώσουμε, να δώσουμε το, το, το, το το ε, οποίο θέλουμε ή στην Ευρωπαϊκή Χρονιά να εμπλέξουμε τις τοπικές περιφερειακές αρχές σε κάθε επίπεδο και έτσι εδώ πέρα να αντικατοπτρίσει αυτές τις δράσεις μας το θέμα του ότι είναι αυθεντική η λύση η Ευρώπη για τα 8 δις των, των, των, των, των ατόμων που γίνονται σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Επίσης να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη δέσμευση του με αυτά τα 5 εκατομμύρια τα οποία ανέφερε η Αντιγόνη, και το, το ετώνησε και η πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι αυτό ε, ε, είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Οικονομία, τον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνουν τέτοιε οικονομίε. Και επίση μου ανέφεραν ότι υπάρχει θέμα ε, εγκυρότητο αυτή τη τροπολογία. Να το δούμε αυτό, γιατί έχουμε την απόφαση του 2012 που περιέχει ακριβώ την ίδια διάταξη, ταυτόσημη. Δεν καταλαβαίνω γιατί επομένω η δική μα τροπολογία δεν είναι παραδεκτή. Επίσης, ε, το, το θέμα δεν είναι το θέμα, είναι ότι είναι, είναι πολύ σημαντική. Επομένω, φέτος θα πρέπει ε, ε το τα οποία κάνουμε φέτο να έχουν προκοδοθεί κατάλληλα, ούτω ώστε να, μπορούν, να μπορεί η προκοδότηση να βρίσκεται στο ύψο των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Επόμενο. Η επόμενη μάλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου ε, τους, τον, του, την εισηγήτρια ή τους εισηγητές, γιατί εκάλυψε ένα σωρό προτάσεις που είχαμε διάφορες εξημών. Επίσης πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ ως επιτοπλίστων με όσα είπε η Ναταλή Γκρισμπέκ ε, και όσα είπε για τον προπολογισμό. Ξέρετε και εγώ έχω την ίδια τροπολογία καταθέσει. Είχαμε εμπλακεί πάλι στην προηγούμενη τέτοια ευρωπαϊκή χρονιά, είχαμε ζητήσει αύξηση προοικοδότηση και αυτό μου φαίνεται κάπω περίεργο το ότι άπαξ και έχουμε με τέτοιο έτος Ευρωπαίου πολίτη να κάθομαστε και να μην έχουμε, μην έχουμε ε, μια παρική προοικοδότηση, να έχουμε τον το πιο χαμηλό προπολισμό που έχει ποτέ προβλεφθεί για τέτοια ε, για χρονιάς. Επομένως θα πρέπει να δούμε το ότι θα πρέπει να εστιάσουμε προσοχή μας στον Ευρωπαίο, στον Ευρωπαίο πολίτη. Δεν νομίζω ότι έχει να μας πει τίποτε παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να μην το ξέρουμε. Και η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής νομίζω ότι θα πρέπει περισσότερο να αντικατοπτρίζει αυτό το ενδιαφέρον για τον πολίτη. Αν αυτό γινόταν τότε και εμείς θα είχαμε και εγώ τροπολογίε. Πάντω, βλέπω μια και που είμαι συγκεντρική και εντροπή πολιτικών θεμάτων, ότι αυτό το οποίο μας λέει η Επιτροπή και το Συμβούλιο, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει μεταβληθεί καθόλου μετά από τόσες και τόσες μέρες που τα συζητούμε. Άρα θα πρέπει και εμείς δυναμικότερα να προβάλλουμε τις απόψεις μας για τους Ευρωπαίους. Και ακριβώς λόγω της ιδιότητάς μας ξέρουμε τι ζητάει ο Ευρωπαίος. Κυρίως θα πρέπει αυτό να είναι σημαντικό μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Να προσπαθήσουμε επομένω να, να σταματήσουμε να λέμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Επίσης, να σας αναφέρω και κάτι άλλο. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε στην προηγούμενη συζήτηση. Όπως σας είπα, είμαι συγγήτρια και της Πολιτικής Επιτροπής. Οπότε, για την εκπαίδευση παιδεία προς τους Ευρωπαίους υπάρχει το θέμα του πώς θα καλύψουμε και τους νέους και πώς θα εμπλέξουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτούς και τους ανήλικους. θα πρέπει κανείς να συνειδητοποιεί τους Ευρωπαίους πολίτες όσο γίνεται νωρίτερα. Νομίζω ότι όλες ήθελα να σας πω, σας τα είπα. Mr. Bronx, now your turn. Thank you. When I first heard that 2013... Όταν η πρώτη φορά άκουσα το 2013 θα ήταν η χρονιά του Ευρωπαίου πολίτη, λέει ο κύριος Μπρόνς, κάπως άρχισα να αισιοδοξώ. Ωραία, 2013, και να αργήσει λίγο θα μεγάλα. Όχι, έκανα λάθο, γιατί αυτό αναβάλλεται συνέχεια, συνέχεια μετατίθεται. Λέει εδώ πέρα η συγγήτρια κάποια θέματα για τη στήκη του Μαστρίχ και είπε ότι τότε θεσπίστηκε η ιδιότητα αυτή, ούτω ώστε να αναδείξει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και επίσης την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Βέβαια. Άλλο ηθαγένεια και άλλο ηθαγένεια Ευρωπαίου πολίτη. Στην κρίκο είναι κάποιο κριτήριο σαν τον τόπο γεννήσεως ή την καταγωγή. Ενώ τώρα εδώ έχουμε θέματα υποκειμενικά. Ταυτότητα, εθνικότητα εδώ, μπερδεύονται. Όχι, η εθνικότητα θα πρέπει να είναι η ιδιότητα του, του πολίτη. Άλλο ταυτότητα και άλλο εθνικότητα. Τι γίνεται όμως με αυτή την ιδιότητα του πολίτη. Κοινή ιστορία, κοινός πολιτισμός, αυτά είναι κοινά μας. Όπως είναι κοινή και η πόλεμη του ενός εναντίον του άλλου. Αυτά όλα είναι προέκταση της εθνικότητας, αλλά και στενότερα αυτής, όχι το αντίστροφο. Πάντοτε η εθνικότητα, η καταγωγή κατήσχε. Πρόκειται για εφευρήματα αυθαίρετα δεν προκρίνουν κανένα είδου ταυτότητα, κοινή αντίληψη και τέτοια. Το αντίθετο. Όχι, πρόκειται για τους προγόνους μας, για τον πολιτισμό κλπ. κλπ. Όλα αυτά δεν γίνονται να είναι σε επίπεδο Ευρώπης. Η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη δεν αρκεί για να φτάσουν στην κοινή ταυτότητα. Τι ενδέχονται κάποιοι τριτοκοσμικοί και ευθύνονται και αυτοί για το ότι ολένα και έχουμε δημορφικό πρόβλημα. Οπότε έτσι και η περιορισμένη αίσθηση του ανήκειν που υπήρχε και αυτή καταπίπτει. Τόσο σαν αφορά την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Καλά τώρα, τώρα να δίνουμε τόσο πολύ σημασία σε αυτό, σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε τίποτα να κάνουμε, θέλουμε να κυκλοφορούμε γύρω-γύρω, αυτό δεν ισχύει. Όμως θα πρέπει τελικά να λάβουμε υπόψη ότι αυτό εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις. Πώς θα κερδίσουν περισσότερο. Άλλο ενιαία αγορά και άλλο που μένουν σε ιδιότητα πολίτη κλπ. κλπ. Το ευρωπαίο, ευρωπαϊκό όραμα είναι επιχειρηματικό. Άλλο οικονομία, άλλο άνθρωπος. Και δεν πρέπει ποτέ ο άνθρωπος να θυσιάζεται επομένω στο βωμό τη δημιουργία ηλική ευημερίας. Έχουμε τις ευρωεκλογέ, έχουμε τις ε, δημοτικές και κοινωτικέ εκλογέ. και θα πρέπει εδώ να μην ξεχνούμε ότι το πάνω χέρι το έχει σε αυτές τις εκλογές ο λαός και όχι κάποιος που βρίσκεται κάπου και τα κανονίζει όλα. Ο Δήμος, ο Δήμος, ο κόσμος Επομένως όλα αυτά το οποία το Βενιδιώδιο του Ευρωπαίου Πολίτη είναι αυθαίρετα, είναι ένα αυθαίρετο συμπίλημα που προσπαθούν να φτιάξουν. Μακίνταρ. Εγώ διαρωτώ με αν ο χρονισμός είναι ο σωστός για το να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Χρονιά πολίτη ηθαγένεια το 2013. Πρέπει να ομολογήσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε και αυτή αντίστοιχες ανησυχίες όταν αναφέρθηκε στη ποσά τα οποία έχουν δαπανηθεί. Υπάρχουν προβλήματα συγκυρίας, υπάρχουν προβλήματα σε χώρες όπως η Ελλάδα, υπάρχουν υψηλά επίπεδα ανεργία σε χώρες όπως η Πορτογαλία και πολλοί θα πίστευαν ε, ότι δεν υπάρχει χώρος και δυνατότητα σε αυτή τη φάση για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα ή να πείσουμε τους πολίτες να νιώσουν ότι είναι πολίτες της Ένωσης. Αυτό δεν δικαιολογείται. Υπάρχει κάτι όμως το οποίο με θλίβει, πραγματικά με θλίβει είναι ότι η έκθεση αυτή και πολλές από τις τροπολογίες συστηματικά αναφέρονται στα δικαιώματα των πολιτών. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στα καθήκοντα των πολιτών. Τα δικαιώματα και τα καθήκοντα είναι οι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος, του νομίσματος της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη. Έχεις το δικαίωμα να εκλέγεις, αλλά έχεις και το δικαίωμα και την ευθύνη του να εκλέγεις. Η δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες λοιπόν στον πολίτη, ακριβώς επειδή είναι πολίτης. Να αναφερθώ σε έναν γνωστό, ε, τον Edmund Burke, ο οποίος ήταν ε, ένας ε, Ιρλανδός του 18ου αιώνα, πέρασε πολλά χρόνια στην Κάτω Βουλή. Στην ουσία θεωρείται ο φιλοσοφικός, θα έλεγα, ηγέτης ε, του συντηρητισμού του Βρετανικού σήμερα. Είπε ότι το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι οι καλοί και σωστοί άνθρωποι να μην κάνουν τίποτα, να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ενώ το ζωτικό στην δημοκρατία είναι ο πολίτης να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Όχι μόνο δικαιώματα λοιπόν αλλά και καθήκοντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Σντάνοκα, αν ακούσαμε καλά. Ναι, η κυρία Σντάνοκα. Υποστηρίζουμε τις ιδέες που περιλαμβάνονται και στις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί από πλευρά της πολιτικής μου ομάδας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα θέματα τα οποία φύγουν οι τροπολογίες αυτές θα ήθελα επίσης να θέσω ένα ερώτημα στην κυρία Παπαδοπούλου και στους εκπροσώπους περισσότερο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αλλαγή του τίτλου. Δεν μιλάω για τυπικό θέμα, αλλά θέμα έννοιας. Τι ακριβώς θέλουμε να πούμε εμείς στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας την οποία κάνουμε για τη χρονιά αυτή για το έτος του πολίτη ή για το έτος της ηθαγένειας. Όπως έχω ήδη πει μέχρι τώρα σε προηγούμενες συζητήσεις, υποστηρίζουμε με την προσπάθεια, αλλά νομίζουμε ότι με την αλλαγή του τίτλου θα υπάρξει μια αλλαγή κατεύθυνσης. Θα εμείνουμε περισσότερο στην ιδέα της ηθαγένειας και στο τι σημαίνει η ηθαγένεια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το θετικό, είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει προσθετικά σε όλους οι οποίοι ζουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τους κατοίκους και παραμένοντες γενικότερα στα εδάφη, της, ε, στους μόνιμους ε, κατοίκους εδώ τίθεται και το θέμα της διπλής ηθαγένειας, τίθεται επίσης το θέμα της εναρμόνισης των νομοθετικών ρυθμίσεων, Νομίζω ότι η πρόταση αυτή λοιπόν είναι πιο θετική. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε και τις γνωμοδοτήσεις της ε, ε, Επιτροπής ε, Αναφορών και ο κύριος Σταυρακάκης δεν είχε ακούσει για την πρόταση για την αλλαγή του τίτλου. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια, μιας και υπάρχουν και τέσσερις γνωμοδοτήσεις, Πώς θα προχωρήσετε με την πρότασή σας αυτή για την αλλαγή του τίτλου. Τι ακριβώς στοχεύετε μεθοδολογικά να κάνετε για να πετύχει η προσπάθεια, την οποία βρίσκω καλή και πρέπει να πετύχει. Ευχαριστώ κυρία Σντάνοκα. Η κυρία Παπαδοπούλου τώρα ακούσατε πολλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω απαντώντας τελευταία ερώτηση. Ο λόγος για τον οποίο ζητούμε την αλλαγή του τίτλου είναι ότι αρχικά αυτό είχε ζητήσει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου του 2010. Το δέτος αυτό χαιρετίζει την 20η επέτειο από την συμπερίληψη συνθήκη της, ε, του Μάστερ του 1993 της έννοιας Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Ο τίτλος λοιπόν αυτός, αντί να μιλούμε για Ευρωπαϊκότητα του πολίτη ε, έχει σαν στόχο να προβάλλουμε όλα αυτά τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες, τα δικαιώματά τους, τον τρόπο να προστατευτούν τα δικαιώματα αυτά, να γνωρίζει ο πολίτης τα δικαιώματά του, τι μηχανισμούς έχουμε στην Ένωση να τους υποστηρίξουμε και πράγματι σε περίοδο οικονομικής κρίσης πολλές ανησυχίες και ερωτήματα που απασχολούν τον πολίτη ε, καλούν να δοθούν εξηγήσεις για το τι σημαίνει η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Συμφωνώ το όντι ότι δεν πρόκειται μόνο για δικαιώματα, αλλά και για ευθύνες. Υπόθηκε νωρίτερα ότι είναι πολύ σημαντικό και οι δύο πτυχές να υπογραμμιστούν Οι μετρήσει του Ευρωβαρομέτρου όντω έδειξαν ότι υπάρχει επικρατή άγνοια που τι σημαίνει η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Μερικές φορές ο πολίτη θεωρεί ότι αυτό του ε, τον επιφορτίζει με περισσότερες ευθύνες από δικαιώματα. Και όντω, λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο πολίτη να συμμετέχει Υπογραμμίζουμε ιδιαιτέρως στην έκθεσή μας ότι η συμμετοχική δημοκρατία θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των μελημάτων μας και ιδιαίτερα θέλουμε να υπογραμμίσουμε και να τονίσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία στηρίζεται στην κοινή ιστορία, τον κοινό πολιτισμό, δεν μπορεί να είναι τεχνητή. Και έτσι, διευρύνοντα τα δικαιώματα αυτά που δεν σημαίνουν μόνο ότι μπορεί κανείς να πάει και να εγκατασταθεί σε ένα άλλο κράτος μέλο, αλλά ότι μπορεί να ψηφίσει και να εκλεγεί, ότι μπορεί να κάνει αναφορά στο κοινοβούλιο ή στον διαμεσολαβητή, ότι μπορεί να συζητήσει την εξέλιξη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση με άλλου συμπολίτε του πολίτη της Ακριβώς ε, νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζει τι συνεπαγόνται τα δικαιώματά του. Και όπω είπε και η Επιτροπή, πρέπει να επικεντρωθούμε στον άνθρωπο και όχι μόνο σε αρχέ και διαδικασίε μόνο. Για να το πράξουμε όμω αυτό, θα πρέπει το όντι να έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότερο, περισσότερα κονδύλια, γιατί είναι τόσο περιορισμένος ο προϋπολογισμός που εν τέλει θα επιβληθούν μόνο άνωθεν προσδιοριζόμενες πολιτικές και δεν θα υπάρχει περιθώριο για ε, συμμετοχή και συμβολή του πολίτη στην ε, χρονιά αυτή. Όντω, με απασχολεί πολύ αυτό. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλογιστεί τι δυνατότητε θα μπορούσε να έχει για να ενισχύσει τον προπολογισμό. Εμείς ε, στοχεύουμε στην επίτευξη Συμφωνία στο χύτερο δυνατό μεταξύ Επιτροπής και με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να υλοποιηθεί το ευρωπαϊκό έτος. Δεν είναι σαφές για μένα εάν το, όντως, το όντι το Κοινοβούλιο στηρίζει την γνωμοδότησή μου, διότι η πρώτη δήλωση που άκουσα από εκπρόσωπο του Συμβουλίου ήταν το Συμβούλιο υποστηρίζει πλήρως τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ίσονε τροποποιήσει. Εγώ όμω έχω, επιβα... έχω επισημάνει συγκεκριμένα και ζωτική σημασία στήματα όπω την άξιση του προπολογισμού, την αλλαγή του τίτλου. Θεωρούμε ότι είναι η θαγένεια καλύτερο η έννοια από τη λέξη πολίτης απλώς και θα θέλαμε περαιτέρω διευκρινήσει των θέσεων του Συμβουλίου. Εν τέλει, και αφού άκουσα τα όσα είπε η κυρία Γκρίσπερ και η κυρία Βλέζια, θα ήθελα να πω ότι και εγώ συμφωνώ πως όντως θα πρέπει ως κοινοβούλιο να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ενισχύσουμε την ε, ε, συνειδητοποίηση πλευρά του πολίτη, του μηνύματος, ε, του, της εμβέλειας, του δυναμικού. Γιατί ναι, λόγω αυτής της μεγάλης οικονομικής κρίσης διαπιστώνεται απουσία ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης. Υπάρχουν χώρες οι οποίες γνωρίζουν τεράστια προβλήματα οικονομικά και διαρωτώνται εάν ήρθε η ώρα πλέον ο πολίτης τους να αναζητήσει άλλη μοίρα και να φύγει από τον Νότο στην κεντρική, στη Βόρεια Ευρώπη για να βρει θέσεις εργασίας ή αν μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να αναπτύξουμε στις χώρες μέλη ε, τις ε, συνθήκες εργασίας που, που χρειάζεται. Είτε δηλαδή κάποιος πάει για να δουλέψει, είτε για να σπουδάσει, είτε για να βρει συνθήκες διαβίωσης ε, διαφορετικές σε μια άλλη χώρα μέλος, θα πρέπει να έχει πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων του, που των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, χωρίς την ιαδήποτε ή παραμικρή διάκριση. Αυτά είναι τα ερωτηματικά που μας απασχολούν, αυτά είναι τα ερωτηματικά που καλούν οι απαντήσεις και τώρα στη χρονιά αυτή την Ευρωπαϊκή ήρθε η ώρα να δώσουμε απαντήσεις πιστεύω και να ενισχύσουμε την ε, ευαισθητοποίηση, την ε, συνείδηση του πολίτη για το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Θαγένεια, τι θα φέρει αυτό το έτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδοπούλου. Σας ακούσαμε, ακούσαμε τα επιχειρήματά σας και τα επιχειρήματα των, κρατών μελών, των ε, συναδέλφων μας των μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο μετά τη συζήτηση αυτή έχουν κάτι να προσθέσουν. Σύντομα, όχι. Σας ευχαριστώ. Όχι και τότε προχωράμε. Ακούσαμε τους συναδέλφους, την κυρία Παπαδοπούλου Σίγητρια Πρέπει ως εκ τούτου να προσδιορίσουμε μια προκαταρκτική ψηφοφορία για τις 8 Μαΐου, όπως έχει ζητήσει η εισηγήτρια, να έρθει λίγο πιο νωρίς δηλαδή ψηφοφορία, έτσι δεν είναι τις πρώτες ημέρες του, μάλλον να πάει αργότερα, τις πρώτες ημέρες του Μαΐου αντί του Απριλίου. Ας κοιτάξουμε τώρα το έκθεση του κυρίου Κορνέλης Δε Γιόγκ, του ποινικού δικαίου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έκθεση. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εδώ, εναρμόνιση του, της έννοιας του εγκλήματος ή του αδικήματος, την ανάπτυξη χώρου δικαιοσύνης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα αφού η, Ευρωπαϊκή, η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησε ζήτημα ευρωπαϊκό το χώρο της δικαιοσύνης, χώρο τομέα δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής και άρα στόχο ο οποίος είναι και στόχος μεγάλος, μεγάλη πρόκληση που θα πρέπει να επιτευχθεί και με την βελτίωση της ποιότητας και τη αποτελεσματικότητα τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στον χώρο του ποινικού δικαίου, που ταυτόχρονα θα σημαίνει ευθυγράμμιση ε, και τήρηση και των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπω τα περιγράφει όχι μόνο ο Ευρωπαϊκό Χάρτη, αλλά και όπω τα ορίζουν οι παραδόσεις, ε, το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο άλλωστε μία συνάντηση που είχε θέσει υπό την αιγύδα τη η Επιτροπή μα στα τέλη του 2011 το Δεκέμβριο συγκεκριμένα, ε, οδήγησε στην απόφαση για διατύπωση έκθεσης ιδία πρωτοβουλίας από τον κύριο De Jong, συντάκτη, ο οποίο έρχεται τώρα να μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθέσεω του. Έχετε το λόγο κύριε De Jong. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καιρό τώρα Καιρό τώρα έχουμε κάνει, έχει, καιρός τώρα έχει περάσει από την τελευταία συνεδρία με τους κοιόδους ηγητές. Είχα ετοιμάσει το σχέδιο. Ε, πρέπει να πω όμως ότι η συνάντηση που διεξήχθη ήταν και πάρα πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα δε η ακρόαση, όπου προσκαλέσαμε ερευνητές πανεπιστημιακούς για να ακούσουμε τις απόψεις τους. Εγώ είχα επαφές και με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, της Επιτροπής, των κρατών μελών, με εκπροσώπους των πανεπιστημίων. Από τη συζήτηση αυτή λοιπόν, από την ακρόαση αυτή, απορρέει το εξή μήνυμα. Ότι στο ποινικό δίκαιο πρέπει κανείς να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή ε, και σύνεση τόσο στο εθνικό δίκαιο όσο και στο ευρωπαϊκό, πολλομάλλον δεν στο ευρωπαϊκό, γιατί το παραμικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντικά προβλήματα. Αν ακούει κανεί τι εφημερίδε ή το ραδιόφωνο ότι ε, εκδηλώνονται κάποιε ε, ε, πράξεις ιδιαίτερα εντυπωσιακές μπορεί να έχει ως αυθόρμητη αντίδραση την επιβολή μια νέα κύρωση μέσω του ποινικού δικαίου, θεωρώντα ότι μια τέτοια διάταξη μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα. Ωστόσο, όλοι οι ειδικοί με του οποίου συνομίλησα με προειδοποιούν ότι αυτό είναι ασφαλμένη επιλογή. Το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στο πλαίσιο ενό ε, ενθουσιασμού ε, νομοθετικού ε, που θα οδηγούσε σε πολλαπλασιασμό των χαρακτηρισμών και των, των πράξεων και των κυρώσεων, του χαρακτηρισμού των πράξεων και των κυρώσεων. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια σαφής ε, παράδοση στην Ευρώπη, διαφορετική στα κράτη-μέλη, η οποία έχει οδηγήσει σε επιλογές διαφορετικές πολλές φορές, Φερρυπίν, στο θέμα της ευθανασίας και το κάθε κράτος έχει το δικό του μερίδιο, τη δική του ε, τοποθέτηση σε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία δεν χωρεί εναρμόνιση. Αυτό προσπαθώ να αντικατοπτρίσω και στην έκθεσή μου. Ότι πρέπει οι ιδιαιτερότητες κάθε κράτους, κάθε χώρας να παραμείνουν πάντα μέσα στο πλαίσιο βέβαια των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να παραμείνει ενισχύ. Και μόνο εάν υπάρχει ανάγκη θα ε, καταφεύγουμε στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο. Ε, έτσι λοιπόν πέραν αυτών των δηλώσεων και διακηρύξεων, εξέτασα το πώς θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τα λειτουργικά στοιχεία του δικαίου αυτού. Ε, πώς θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε τη συμμετοχή όλων των παραγόντων στη διαμόρφωση του δικαίου αυτού. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η, η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών δεν έχει μονοπόλιο στη συζήτηση αυτή, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αρμοδιότητα σε κάθε τομέα ε, της πολιτικής ε, που χαράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, λαμβάνει αποφάσεις στο όνομα των πάντων. Ξεχνάμε ότι ακόμα και στον τομέα του περιβάλλοντος πλέον έχει επιφυλοχωρήσει το ποινικό δίκαιο. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να διατηρούμε μια γραμμή ενιαία στο ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ως προς την προσέγγιση των ποινικών θεμάτων. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και όπως είπα επαγρυπνώντας ώστε, ε, ώστε να έχουμε σωστή διατύπωση των όρων όταν πρόκειται για ένα ποινικό αδίκημα. Ένας, ε, μια υπηρεσία συντονισμού για το ποινικό δίκαιο επίσης που έχει προβλεφθεί θα μπορούσε να αποτελέσει μια χρήσιμη μονάδα στο βαθμό που δεν θα ασχοληθεί με μια συγκεκριμένη κατηγορία δικημάτων, αλλά που όντως θα επιτελέσει το έργο της ως ε, μονάδα συντονισμού των ε, ε, ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το ποινικό δίκαιο. Τώρα έχει έρθει η ώρα λοιπόν, αφού εξέτασαν το ζήτημα και η Επιτροπή και το Συμβούλιο, να διατυπώσει και το Κοινοβούλιο τη θέση του. μέσα σε ένα κείμενο που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό, ε, συνεπές και ακριβές διατύπωσή του. Με στόχο να ευθυγραμμιστούν στις ίδιες τοποθετήσεις όλα τα θεσμικά όργανα. Πρόεδρε, δεν θα πω περισσότερο. Υπάρχει μια προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών που έχει οριστεί για το Μάρτιο με ψηφοφορία στις 12 Απριλίου στην Επιτροπή μας. Γι' αυτό λοιπόν σταματάω εδώ για να ακούσω και τις αντιδράσεις των συναδέλφων. Ευχαριστούμε κύριε Ντεγιόνγκ. Η Επιτροπή νομίζω θέλει να συμβάλλει στη συζήτηση από πλευρά τη. Έχουμε κάποιον εκπρόσωπο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Η έκθεση αυτή έρχεται σε σωστό χρόνο. Είναι συμβατή με την ανακοίνωση που ε, εκδώσαμε τον μήνα Σεπτέμβριο Υπάρχει υψηλό επίπεδο συμφωνίας με το δικό μας κείμενο και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απλά θα πούμε ότι προσβλέπουμε σε μια καλύτερη διοργανική συνεργασία επί τη βάση της προτάσεως αυτής. Δεν θα κάνω ε, σε αυτή τη φάση παρατηρήσεις επί των λεπτομεριών. Καλώς. Α, κύριος Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή, ο οποίος στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα αυτό μας προσφέρει ε, μία βάση εργασίας. Έχω μια σειρά ίσονος σημασία ίσων σημασια όπου θεωρώ ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε και ιδιαίτερα στο στρατολογική σκέψη Έλα. ΙΒ δηλαδή. Θα ήθελα μία πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση για το πώς βλέπει να διαμορφώνεται αυτή η ιδέα. Στο ΙΓ μπορούμε να έχουμε ενδεχομένως ανάγκη για διακυβερνητική συμφωνία ή μήπως μπορούμε να πούμε ότι όποιος αναλαμβάνει την εκπόνηση αυτού του έργου θα βρίσκει και τη σχετική λύση. Στο δε σημείο 2, στο γερμανικό τουλάχιστον κείμενο όπως το βλέπω, γίνεται λόγος για ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία. Πραγματικά λέει το ελληνικό κείμενο. Θα ήθελα αυτό να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Στα δε σημεία 8 και 10, στην περαιτέρω διαδικασία, θα ήθελα ε, να συζητήσουμε την ενδεχόμενη ε, δημιουργία νέων διοικητικών μονάδων. Είναι ανάγκη και είναι όντως πρακτικά εφαρμόσιμο αυτό το οποίο ζητεί ιδιαίτερα το σημείο 8 δεν είναι υπερβολικό να απαιτούμε τη θέσπιση νέου χαρτοφυλακίου επιτρόπου για ποινικό δίκαιο και δεν θα ήταν και αντιπαραγωγική μια τέτοια ιδέα. μου ότι αν ένα επίτροπο έχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, προσπαθεί πάντοτε να το εμπλουτίσει με μια σειρά από νέε διατάξει ε, και άρα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξελίξει στον χώρο του ποινικού δικαίου που ίσω ε, να είναι αμφίβολων αποτελεσμάτων και νομιμότητας και πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέος επίτροπος, νέα υπηρεσία, γενικές διευθύνσεις και γενικά όλος ο μηχανισμός που συνεπάγεται αυτό θα ήταν μάλλον εσφαλμένη λύση. Ο επίτροπος ή η επίτροπος που έχει αρμοδιότητα γενικά για την ομοθεσία θα μπορούσε να αναλάβει και το χαρτοφυλάκιο του ποινικού δικαίου και εσωτερικά να γίνει κατανομή ενδεχομένω με πολύ μεγάλη προσοχή φυσικά. Αλλά νέο χαρτοφυλάκιο επιτρόπου όχι δεν θεωρώ ότι χρειάζεται και μάλιστα του αντίον θεωρώ ότι θα ήταν και αντιπαραγωγική επιλογή. Στο σημείο 11 θετικά κρίνω το ότι ζητούμε την ενίσχυση της νομικής υπηρεσίας Εν γέννη θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό, διότι και άλλα κοινοβούλια έχουν νομική υπηρεσία. Εμείς πρέπει να περνάμε από το Προεδρείο πάντοτε για την υπόθεση αυτή. Έτσι λοιπόν νομίζω θα ήταν καλό να επισημάνουμε ότι η νομική υπηρεσία χρειάζεται ουσιαστικά να ενισχυθεί. Και στο σημείο 3 εν τέλει, εκεί που λέτε ότι να γνωρίζονται οι άλλε γενικέ αρχέ που διέπουν το ποινικό δίκαιο, Αυτέ οι γενικές αρχές ξέρω ότι βέβαια μας περιορίζει η έκταση που έχει οριστεί ε, εκ των προτέρων για κάθε έκθεση, αλλά θα πρέπει ίσω να είμαστε πιο αναλυτικοί ως προς τις ε, γενικές αρχές. Ξέρω ότι δεν είναι διεξοδικός ο κατάλογος, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάποιες ακόμη πέραν αυτών των τριών που καταγράφονται, διότι δεν επαρκούν, πιστεύω, οι τρεις μόνο γενικές αρχές ε, για να εξαντλήσουν την έννοια του ποινικού δικαίου. Πρέπει να προσθέσουμε μερικά στοιχεία ακόμη. Ευχαριστώ. Βαρόνι Λάτφορντ. Σειρά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς τον κύριο Ντεγιόν. Η έκθεσή του είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Πράγματι απαιτείται να συντάξουμε ένα κείμενο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο που να προσθέτει αξία. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση απλά να ανακατευτούμε στις αλλαγές του ποινικού δικαίου των κρατών μελών. Το θέμα αυτό πολιτικά μάλιστα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Το θέμα τίθεται εν πάση περιπτώσει και πολιτικά για τους γνωστούς λόγους. Ε, πέραν αυτού όμως υπάρχει θα έλεγα στήριξη της κοινή γνώμης ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι βασικές προτεραιότητες που θέλει ο κόσμος να κάνει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, περιέχουν και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με συντονισμένο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν στήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα με σωστό τρόπο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν να κατανοήσουμε τις αρχές όμως της αναλογίας και της επικουρικότητας όπως μας προτείνει ο κύριος Ντε Ιόγκ. Απαιτούνται βέβαια και κοινά διαδικαστικά νομικά βήματα μια θα έλεγα <clears throat> κοινή νομική ρύθμιση χωρίς να καλύπτει την μεθοδολογία τη οποία πρέπει να ακολουθείτε κάθε φορά δεν έχει νόημα. Πρέπει να υπάρξει μια, ένα κοινό στάδιο εδώ. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς τις σωστές ρυθμίσεις αλλά είναι και δύσκολο να επιλέξει τις σωστές πρακτικές χωρίς να επηρεάσει κανείς την οργάνωση των εθνικών, των εσωτερικών θα έλεγα ποινικών συστημάτων. Τίθεται εδώ το θέμα του ποινών, τίθεται το θέμα των κρατήσεων και δημιουργούμε θέλοντας ή όχι θα έλεγα προκλήσεις σχετικά με κάποια ε, θέματα πολιτικά ευαίσθητα όπως οι ελάχιστες ή οι μέγιστες ε, ε, επιτρεπόμενες ποινές κτλ. Απαιτείται λοιπόν μεγαλύτερη θα έλεγα απόδειξη από πλευράς μας της ικανότητάς μας να λειτουργήσουμε με τρόπο συνεκτικό σε σχέση με το ποινικό δίκαιο απαιτείται καλύτερο συντονισμός ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Συμφωνώ με τον ομιλητή που είπε ότι δεν πρέπει, τον εισηγητή που, δεν είπε ότι, που δεν πρέπει να υπάρξει μια νέα γραφειοκρατία η οποία να επιβαρύνει την κατάσταση και νομίζω ότι και η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε ένας επίτροπος να ασχολείται με τα θέματα τα ποινικά είναι κάτι το σωστό. Βέβαια ε, όλα αυτά χρήζουν περαιτέρω συζητήσεων να δούμε σαν παράδειγμα χρειάζεται μια εσωτερική διοργανική συμφωνία πριν περάσουμε σε αυτή τη φάση. Πάντως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ότι στα πλαίσια της συγγραφής της νομοθεσίας αυτής γύρω από τον ποινικό χώρο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους ενδιαφερομένους και εμπλεκομένους εμπειρογνώμονες, εθνικά κοινοβούλια, δικηγορικούς συλλόγους, Eurojust, κοινωνία των πολιτών, όλους αυτούς οι οποίοι θα, τους οποίους αφορά η προσπάθειά μας. Επίσης θα πρέπει να ακολουθήσουμε και τις οδηγίες της νομικής μας υπηρεσίας, η οποία θα είναι χρήσιμο να μας συμβουλεύει και στα πλαίσια της διατύπωσης των νομοθετικών μας προτάσεων, ήδη ίσως να το κάνουν. Εγώ όμως προσωπικά θα ήθελα να πω ότι δεν, δεν θα έλεγα νιώθω πολύ καλά γιατί δεν έχω τη στήριξη ενός κοινοβουλευτικού συντάκτη από πλευράς διοικητικής της γραμματείας του Κοινοβουλίου εννοώ κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι για τις επιπτώσεις των νομοθετικών μας προτάσεων. Κάτι τέτοιο αντίθετα συμβαίνει στην Αγγλία. Θα πρέπει λοιπόν να έρθουμε σε επαφή όχι μόνο με τα υπόλοιπα όργανα αλλά και με τους άλλους εμπειρογνώμονες του θέματος. Χρειάζεται λοιπόν να οικοδομήσουμε και να συμπεριλάβουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα στις νομοθετικές μας ρυθμίσεις γιατί γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη φάση μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα και έχουμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, κάτι το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα, αλλά τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα έπρεπε να μας απασχολήσουν περισσότερο. Ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει εξελιχθεί με αρκετά χαμηλή ταχύτητα, είναι η αναθεώρηση των μέσων τα οποία ψηφίζουμε. Εμείς ε, έχουμε αρκετό καιρό τώρα θα έλεγα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Έχουμε αρκετές αξιολογήσεις αλλά σε σχέση με την εντολή, την ανακριτική, την ευρωπαϊκή, ε, είναι σαφές ότι θα έπρεπε να μπορέσουμε να δράσουμε πιο γρήγορα σαν Επιτροπή, σαν Συμβούλιο, σαν Κοινοβούλιο, ε, και να μην περιμένουμε 10 χρόνια για να αντιδράσουμε και να δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα. όταν έχουν δημιουργηθεί αρνητικές καταστάσεις από τα κείμενα που έχουμε εμείς ψηφίσει. Εν πάση περιπτώσει, συμπερασματικά, απαιτείται περισσότερο συντονισμός, απαιτείται περισσότερη συνεκτικότητα, όχι μόνο ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, αλλά ανάμεσα σε εμά τα μέτρα που προτείνουμε και τους εμπλεκόμενους στον τομέα αυτό. και θα πρέπει οι νομοθετικές μας ρυθμίσεις να μην παρεμβαίνουν ή να παρεμβαίνουν το κατελάχιστον στις εθνικές νομικές θα έλεγα ρυθμίσεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κλείσουμε τα παραθυράκια τα οποία επιτρέπουν τους, τους αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν τον νόμο σε, σε διασυνοριακό επίπεδο πλέον είναι δύσκολο να επιλέξουμε τον σωστό δρόμο, έχω και εγώ κάποιες τροπολογίες ετοιμάσει και η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών θα πρέπει ίσως να παραταθεί γιατί η επόμενη Δευτέρα για μένα μου φαίνεται πάρα πολύ ε, δύσκολο, ίσως Τετάρτη τουλάχιστον. Ε, δεν είναι πολύ σημαντικές και δεν είναι πάρα πολλές οι τροπολογίες μου αλλά θέλω λίγο χρόνο περισσότερο. Η κυρία Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι αυτό το σχέδιο έκθεσης είναι απαραίτητο και δείχνει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έφερε κάποιες αλλαγές στα πλαίσια των οποίων ενισχύει το ρόλο του Κοινοβουλίου και έχει το Κοινοβούλιο τη συναπόφαση σε αρκετούς τομείς. Εδώ ορίζουμε επίσης με διαφορετικό τρόπο ε, και τις διασυνοριακές ε, ε, ποινικά κολάσιμες ενέργειες σε τομείς όπως η σώματεμπορία, σε τομείς όπως ο ορισμός των κυρώσεων και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία δύσκολα ίσως αντιμετωπίζονται και για τα οποία προβλέπονται είτε διοικητικές είτε ποινικέ κυρώσεις. Α πούμε συζητήσαμε, ακούσαμε σήμερα το πρωί το τι γίνεται σε επίπεδο διοικητικών πράξεων στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος στο διαδίκτυο, στον χώρο. Πρέπει λοιπόν σε επίπεδο κυρώσεων να προχωρήσουμε σε μια πλήρη εναρμόνιση του ποινικού ευρωπαϊκού πλέον δικαίου είναι ένας δρόμος τον οποίο ακολουθούμε. Θα πρέπει και το Συμβούλιο να προχωρήσει. Η ομάδα εργασίας η οποία έχει κάνει δεν έχει ακόμα προχωρήσει. Αν η κάθε χώρα επιμένει να κρατήσει μια πλήρη κυριαρχία στο επίπεδο το ποινικό, ε, τότε τα προβλήματα θα είναι πολλά, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος. Πρέπει να προχωρήσει λοιπόν και η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει προσφέρει όσα περιμέναμε να προσφέρει ή όσα περιμέναμε, όσο περίμενε η Επιτροπή να προσφέρει. Το θέμα δεν είναι να δημιουργήσουμε μια νέα θέση επιτρόπου. Πρέπει όμως να υπάρξει μια, θα έλεγα, ένας προσδιορισμός του πεδίου εδώ, ένα νέο χαρτοφυλάκιο θα έλεγα, το οποίο να ορίζει σωστά το τι σημαίνει εναρμόνιση του ποινικού δικαίου. Πρέπει να γίνουν βήματα προς τα εμπρός, τα βήματα όμως αυτά αφορούν ένα πολύ ευαίσθητο χώρο όπως σωστά τόνισε η κυρία Λάντφορντ και θα πρέπει να υπάρξει κάτι περισσότερο από ένας επίτροπος ή από ε, μια νέα διεύθυνση. Θα πρέπει να υπάρξει ένα επιτρέψει την πραγματική εναρμόνιση. Η εναρμόνιση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα εθνικά ποινικά δίκαια. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση ακόμα. Αντίθετα αυτό το οποίο σημαίνει, όπως είπαν και ορισμένοι πανεπιστημιακοί κατά τη διάρκεια της ακροάσεως η οποία είχε διοργανωθεί στο παρελθόν, θα πρέπει να εναρμονίσουμε κυρίως τους στόχους και τα μέσα που έχουμε για να πετύχουμε τους συγκεκριμένους στόχους. Πρόκειται για θέματα τα οποία είναι θα έλεγα εν πολλής ε, φιλοσοφικά, αλλά ελπίζω η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου να προχωρήσει σύντομα και να επιτρέψει στο Κοινοβούλιο και αυτό να ολοκληρώσει τις προσπάθειές του γιατί υπάρχουν τομείς όπως αυτός στους οποίους δεν έχουμε μπορέσει θα έλεγα να προσφέρουμε όσο θα επιθυμούσαμε γιατί δεν έχουμε ίσως ε, την δυνατότητα να το κάνουμε, όχι δεν είναι θέμα έλλειψης βούλησης. Πέρα λοιπόν από τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου που έχει να παίξει ένα σοβαρό ρόλο, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε και αυτή να δημιουργήσει μια υπηρεσία η οποία να μας διασφαλίσει την από, ε, θα έλεγα, σύνεγγης αντιμετώπιση του προβλήματος. Ευχαριστώ κυρία Λόπες. Ο κύριος Μπρόντς έχει ζητήσει το λόγο, τον έχετε. Εγώ είμαι λίγο σαν το θάνατο και τον εφοριακό, πάντα παρόν. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες στον συγκεκριμένο τομέα. Ίσως είναι, ε, θα έλεγα, η περιγραφή την οποία έκανε ο εισηγητής, μια πραγματικά, θα έλεγα, ε, ανεξάρτητη μορφή επεξεργασίας των θεμάτων. Μίλησε για τα εθνικά χαρακτηριστικά, μίλησε για την ανάγκη να είμαστε επιφυλακτικοί και όχι να προτείνουμε νέες κυρώσεις μόνο και μόνο για να δείχνουμε ότι κάτι κάνουμε. Και συμπερασματικά μετά από τα σχόλια του εισηγήτη είναι να μην προσπαθήσουμε ε, να δημιουργήσουμε εδώ κάποιες ε, νέες δομές αν και φυσικά σαν εισηγητής κατέληξε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Ε, υπάρχουν τομείς αντικοινωνικών συμπεριφορών οι οποίες εκφράζονται θα έλεγα διασυνοριακά. Το θέμα ε, δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο ευρωπαϊκό δίκαιο, το θέμα είναι να συμφωνήσουμε καταρχάς σε επίπεδο απελάσεων, εκδόσεων και ε, συνεργασίας με βάση ε, διμερή και όχι τόσο με τέτοιου είδους υπερεθνικά σώματα όπως το Eurojust. Στο παρελθόν αυτού του είδους τα μέσα που χρησιμοποιούσαμε θα έλεγα οδηγούσε κάποιους κατηγορούμενους να δικάζονται πριν εκδοθούν στη συγκεκριμένη χώρα. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει απόλυτα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κορνέσλησεν Γιάνγκ εσείς τώρα για να καταλήξετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους ε, οι οποίοι έλαβαν το λόγο στο θέμα αυτό πολλές ερωτήσεις που, που σε μένα και τον κύριο Φως. Πιστεύω ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να το απασχολήσει το ζήτημα της διαδικασίας. Πρέπει το θέμα του ποινικού δικαίου να το αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα και σοβαρότητα και να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα στο σημείο 11 της εκθέσεως, όπου γίνεται παραπομπή στην αναφορά μάλλον στην νομική υπηρεσία και λέμε ότι έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, δυνητικά σημαντικό ρόλο επίσης για τον μέλλον κτλ. θα μπορούσε αυτό να εκφραστεί μέσα σε συγκεκριμένες ε, προτάσεις, αλλά μέσα σε μια έκθεση. δεν μπορώ να ζητήσω κάτι πιο ουσιαστικό με πιο σαφείς όρους. Είναι κάτι το οποίο μάλλον στο Προεδρείο είναι από αν κανείς έχει διαφορετικές προτιμήσεις δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε ενδεχομένως με την μορφή μιας τροπολογίας. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα εκκρεμή μέσα στο σχέδιο εκθέσεως που μπορούμε να συζητήσουμε. Τώρα για το ΕΛ και για το κατά πόσον χρειάζεται μια διοργανική συμφωνία ε, ή όργανο. Ε, νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας συντονιστικός ρόλος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστω. Αλλά πάντως, πάντα σε συμφωνία μεταξύ μας. Μην ξεχνάμε ότι ο συντονισμός πάντα ανήκει στο Συμβούλιο. Δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να υπαγορεύει κάθε λεπτομέρεια. Είναι κάτι το οποίο ε, παφείται στο Συμβούλιο. Το αφορά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε και τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τις εσωτερικές διαδικασίες ε, μιας, ενός άλλου θεσμικού οργάνου. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε μέσα σε ένα ψήφισμα. Δεν, μπορούμε, δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε στο θέμα. Οπότε νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να τα δούμε σε μια ομάδα εργασία που να είναι διοργανική και έτσι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιο είδους ε, μνημόνιο κατανόηση, κάποια συμφωνία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάπως να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και αυτό να ε, γίνει εγγράφος και όλος ο κόσμος να τηρήσει τα συμπεφωνημένα. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση του Επιτρόπου, ε, καλό με τον όσον ακούσαμε τους προλαλήσαντες, όχι, όχι, δεν πρόκειται για κάποιον ε, για, για κάποια θέση για καινούργια επιτρόπου. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε αν είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερους προς τον προπολογισμό. Πάντως, εδώ με προβληματίζει το ότι έχουμε τουλάχιστον δύο επιτρόπους που είναι συναρμόδιοι για την έκθεση. Ο καθένας έχει το δικό του γραφείο, τους δικούς του συνεργάτες και οι δύο είναι αρμόδιοι. Αυτό όμως ε, σημαίνει ότι δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί όσον αφορά την διεκπαιρέωση της έκθεσης. Χρειάζεται επομένως συντονισμός πολλής. Το πιο σωστό είναι να υπάρχει ένας επιτρόπος. προσοχή, είναι και θέμα δαπανών, θέμα ποιότητας της νομοθεσίας. Επομένω θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε συνεργασία, πώς μπορούμε να κινηθούμε σε ψηλότερο επίπεδο, στα πλαίσια της Επιτροπής, γι' αυτό θέλει το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Να έχουμε λοιπόν να χειρίζεται το θέμα ένας και μόνο επίτροπος, με τον οποίο να συνομιλούμε, στον οποίο μπορούμε να απευθυνόμαστε, Δηλαδή ο καθένας τελικά ε, έχει αρμοδιότητα για ένα ε, συγκεκριμένο τμήμα του, του, του δικαίου και δεν υπάρχει ένας και μόνο... Τώρα πάμε στην παράγραφη παριθμών 2. Εκεί έχουμε την διάταξη που αφορά το ότι θα πρέπει ε, αυτό ρωτώ κάποια πραγματικά στοιχεία, πραγματικά περιστατικά αν δεν προβούμε σε κάποια εναρμόνιση, τότε μπορεί κάποιος που έχει διαπράξει ποινικό δίκημα να αναζητεί τη χώρα στην οποία θα έχει την ευμενέστερη μεταχείριση, ευμενέστερη ποινική μεταχείριση. Επομένως, θα πρέπει επί βάση πραγματικών περιστατικών να ρυθμίσουμε το θέμα. Άλλωστε μιλούμε για εγκλήματα που έχουν διεθνή φύση. Και άρα έτσι δεν μπορούμε να δώσουμε κάποιο είδου συνεκτικότητα και συνέπεια στην ποινική μεταχείριση. Όλος ο κόσμος αυτό το, το, το αναζητεί. Όμως θα πρέπει η ρύθμιση να είναι στεγανή. Γι' αυτό και αυτή η παράγραφος είναι σημαντική. Α, είχα και κάποια άλλα πράγματα να σας πω. Μισό να, να, να τα δω καλύτερα. Ήδη έχουν φυγεί κάποια θέματα που Α, μάλιστα. Η κυρία Λάτφορντ, η εναρμόνιση είναι θέμα που δεν αφορά αυτή την έκθεση. Βεβαίω και πρέπει να υπάρχουν ελάχιστε ε, εγγύσεις Να μπορούμε έτσι να έχουμε εμπιστοσύνη στο ποινικό μας σύστημα. Αλλιώς αναφύγονται πάρα πολλά προβλήματα. Ε, μιλάμε για τα δικονομικά δικαιώματα εδώ. Και πρέπει να αντιζητηθούν τα κριτήρια επομένω στα πλαίσια των ρυθμίσεων που θέλουμε να κάνουμε στο ποινικό δίκαιο. Αυτά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να αναβάλω την προθεσμία, την καταγγελική ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών. Να προχωρήσουμε στην πιο γρήγορα. Πάντως θα πρέπει να δω τι τροπολογίε υπάρχουν. Είχαμε πάντως μέχρι τώρα θετική συνεργασία και με τον σχεδόν συγητή και πιστεύω ότι ταχαίω θα καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό, σε κάποιο αποτέλεσμα. Πρόεδρος, κύριε Ντεγιόνγκ, αν κατάλαβα σωστά, προτίθεστε να μεταθέσετε την καταληκτική ημερομηνία από 5η Μαρτίου ή ποια ημερομηνία? Στα αγγλικά. Όχι, η 7η Μαρτίου είναι η μόνη η οποία αναφέρθηκε, αν αυτό εξυπηρετεί τον Σκιώδη Συγητή. Ε, εβδόμη 7η Τρίτου, ναι, ναι, 7η Τρίτου σας εξυπηρετεί, ρωτά ο Πρόεδρος. Διότι, μα μου λέει εδώ η γραμματεύς, ότι μέχρι τις 14 μπορούμε να πάμε όσον αφορά την κατάσταση των τροπολογιών. Συμφωνείτε, 14 Τρίτου. Και έτσι δεν διαταράσσεται το χρονοδιάγραμμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την ε, ψηφοφορία, την ψήφιση τέλο πάντων του σχεδίου του κειμένου που ετοίμασε ο σχεδίμας ο κύριος Ντε να γίνει ψηφοφορία μόνο λοιπόν στις 12 Τετάρτου. 12 Τετάρτου η ψήφιση και 14 Τρίτου είναι προθεσμοί για τις τροπολογίες. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ.